Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να αρχίσουμε παρακαλώ. Αν έχετε την καλοσύνη, καθίστε στις θέσεις σας. Σας ευχαριστώ. Σας καλωσορίζω όλους Καταρχάς τον πρόεδρο κύριο Φλαό της ε, Βουλής του Βελγίου με τον οποίον θα συμπροεδρεύσουμε σε αυτήν την ε, κοινή κοινοβουλευτική συνεδρίαση και τον πρόεδρο κύριο Ζουγέ, πρόεδρο ε, της Δημοσιονομικής Αρχής. Ξέρουμε ότι αυτή η περίοδος είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ευρώπη, για τους πολίτες μας που περιμένουν απαντήσεις πάνω στο ερώτημα τι γίνεται στην Ευρώπη. Πώς μπορούμε να ε, τους βοηθήσουμε πώς μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερες θέσεις εργασίας για να ζήσουν μέσα σε ένα πλαίσιο ευημερία, σταθερότητας και ασφάλειας. Η συζήτησή μας σε αυτή τη μεικτή κοινοβουλευτική όλο συνεδρίαση είναι, ε, βασίζεται σε ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που, τους καίνε, που μας καίνε όλους. Το θέμα της συνεδρίασης είναι πέρα από την κρίση πώς μπορεί η Ευρώπη να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις. Ένα πολύ καυτό θέμα. Διανύουμε μία από τις πιο δύσκολες οικονομικές και δημοσιονομικές κρίσεις στην ιστορία μας. Αλλά έχουν ήδη προκύψει ορισμένα συμπεράσματα και ορισμένα μαθήματα. Έχουμε λάβει καταρχάς για την σταθερότητα και πώς να αποφύγουμε παρόμοιες κρίσεις στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό από απόψεως εσωτερικών σχέσεων να αναγνωρίσουμε ότι όταν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ε, ε, δουλεύουν μαζί, συνεργάζονται, μπορούμε να ξεπεράσουμε προσκόμματα. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό στο Κοινοβούλιο ε, και έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχουμε πρόοδο μέσω της υπερψήφισης πολλών νομοθετικών πράξεων με ε, οικονομικό περιεχόμενο. Επίσης έχουμε διαγράψει τη γενική δομή ε, της δημοσιονομικής ε, πειθαρχίας, της λειτουργίας των δημοσιονομικών μέσων. Έχουμε διαμορφώσει μια πολιτική καλύτερου συντονισμού λήψης αποφάσεων έγκαιρα για την αποφυγή κρίσεων μεταξύ των κρατών μελών και επίσης τη λειτουργία ενός πλαισίου αυστηρού, πλαισίου εποπτείας που να επικεντρώνεται στην παρακολούθηση της λειτουργίας των τραπεζών και των αγορών. Έχουμε επίσης υιοθετήσει ε, νομοθεσία για τις επιστολιπτικούς οργανισμούς για την αξιολόγηση των ιδρυμάτων ε, που εγκρίνουν ε, τις πιστώσεις και, και κρίνουν την επιστολιπτική ικανότητα. Επίσης έχουμε καταλήξει σε συμφωνία για τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου εποπτείας για τα hedge funds το οποίο, η οποία πρόταση θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Συμβουλίου και έχουμε επίσης ε, εισαγάγει πάρα πολλά μέτρα ενίσχυσης ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ένα ολόκληρο οικοδόμημα παροχής μικροδανείων τα οποία βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ιδίως σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών προς αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι ένας στυλοβάτη της οικονομίας μας και ένας πολύ σημαντικός παίκτη στην αγορά της Ευρώπης. Θέλουμε λοιπόν να διαμορφώσουμε αυτή την αγορά με μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία. Όσον αφορά τώρα την ε, μελλοντική νομοθεσία, τα μελλοντικά νομοθετικά μέτρα, όπως τα προγραμματίζουμε. Έχουμε αρχίσει να εξετάζουμε άλλους τομείς της οικονομίας αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετούς φακέλους στα χέρια μας που εξετάζονται. Καταρχάς την οικονομική διακυβέρνηση. Το φάκελο της οικονομικής διακυβέρνησης είναι πολύ σημαντικός και ε, από απόψε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικό να εισαγάγουμε κοινοτικά μέτρα, κοινοτικές μεθόδους. Δεν χρειάζονται μόνο η μη οικονομική ένωση ε, αλλά και η νομισματική ένωση. Μην κοιτάμε λοιπόν το ένα σκέλος μόνο της κοινότητας και το οικονομικό και το νομισματικό. Όσον αφορά τώρα την υπερχρέωση, τα swaps και τα παράγωγα, όλα αυτά τα προϊόντα της ε, κερδοσκοπικής, ε, των κερδοσκοπικών συναλλαγών που σε μεγάλο μέρος ήταν τα αίτια της κρίσης, εδώ ε, θα, δημιουργήσουμε μία ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο εγγυάται αποζημιώσει σε περίπτωση παραβάσεως καθηκόντων και νομοθεσιών και για να επανεδρεώσει την αξιοπιστία του πολίτη στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τρίτον, από τη στιγμή που έχουμε καταφέρει να σταθεροποιήσουμε τις αγορές και να αντιμετωπίσουμε μερικά από τα τρέχοντα οικονομικά προβλήματα, θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στη στρατηγική εξόδου από την κρίση, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τις πληγήσεις οικονομίες να βγουν, να ξεπεράσουν αυτή την κρίση, το λεγόμενο exit strategy, δηλαδή μια στρατηγική εξόδου και ανάκαμψης από την κρίση που είναι πολύ πιο ε, σημαντική από την ε, διαχείριση της κρίσης. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε με αυτή τη στρατηγική εξόδου και ανάκαμψης ε, τη δημιουργία δυναμικής ανάπτυξης παραγωγικής ανάπτυξης των χωρών, των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εξέδωσε ένα μια ανακοίνωση την περασμένη εβδομάδα με 15 ε, ε, προτάσεις για το ξεπέρασμα της κρίσης 2011-2012. Η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξε πόσο μπορούμε να συμβάλλουμε εμείς σε αυτή αυτές ε, στην εξέβρεση απαντήσεων στην εσωτερική αγορά, για τα προβλήματα της εσωτερικής αγοράς. Είχαμε με τον αρμόδιο επίτροπο, τον κύριο Μάριο Μόντι, ενδελεχείς και εις βάθος συζητήσεις και αυτή η συνεργασία ήταν πολύ καρποφόρα το 2010. Είμαστε πεπισμένοι ότι για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη μεκροχρόνια ανάπτυξη θα πρέπει να ξεπεράσουμε πάνω από 150 προσκόμματα τα οποία ακόμα υπάρχουν στην ε, εσωτερική αγορά, στην κοινή αγορά και ε, επηρεάζουν την ανάπτυξη. Πρέπει να επιτύχουμε έναν ίδιο ρυθμό ανάπτυξης όπως τότε που είχαμε σχεδιάσει το πρόγραμμα του 1992 της κοινή εσωτερικής αγοράς. Θα θυμόσαστε πάρα πολύ καλά με τι δυναμισμό έχει προχωρήσει αυτό. Επίσης για τα εθνικά κοινοβούλια είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετάχουν στη διαμόρφωση αυτής, αυτού του νομοθετικού πλαισίου. Όταν λέμε νομοθεσία, νομοθετικό πλαίσιο, νομοθετικά μέτρα, μιλάμε για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά χωρίς την συμβολή και τη σύμπραξη των ε, εθνικών κοινοβουλίων δεν θα επιτύχουμε τίποτα. Διότι η εφαρμογή και η ενσωμάτωση του κοινωτικού δικαίου στο εθνικό είναι ίσως ακόμα πιο σημαντική από την αρχική φάση της διαμόρφωσης της νομοθεσίας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η ανάπτυξη και η διατήρηση των σχέσεων με τα εθνικά κοινοβούλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε να λάβετε μέρος σε αυτή την σημαντικότερη ε, συνεδρίαση τη διακοινοβουλευτική και πιστεύω ότι η συνεργασία μας βασίζεται σήμερα αλλά και στο μέλλον πάντοτε δηλαδή θα βασίζεται στην αλληλεγγύη μεταξύ των αρχών αλλά και μεταξύ των πολιτών. Επίσης βασίζεται στην αρχή της ευθύνης, πρέπει όλοι να είμαστε υπεύθυνοι, γιατί είμαστε συνδεδεμένοι μέσω του πλαισίου αλληλεγγύης. Και επίσης, εκτός από την αλληλεγγύη και την ευθύνη, πρέπει να δημιουργούμε, να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικό. Πώς θα βοηθήσουμε τον ανταγωνισμό. Λοιπόν, ο ανταγωνισμός πάντοτε έχει άμεση επίπτωση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και η πρώτη ομάδα εργασίας ακριβώς θα συζητήσει αυτό το θέμα. Τι είδους δηλαδή ανάπτυξη ε, και αγοράς εργασίας προβλέπουμε για την Ευρώπη του αύριο και η ομάδα εργασίας 3 θα ασχοληθεί με το θέμα της, ε, της ευρωπαϊκής κοινή ε, αγοράς και η ομάδα 2 με την οικονομική διακυβέρνηση. Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά μπροστά μας και, αλλά πριν αρχίσουμε τη συζήτηση θα ήθελα να ζητήσω από τον συνάδελφό μου κύριο Αντρέ ε, Φλαχό, Φλαχό πρόεδρο της ε, Βουλής ε, του Βελγίου να λάβει το λόγο και συμπρόεδρο της συνεδριάσεως. σύμφωνα με την αρχή της συμμετοχής για να επανέλθω και σε μια έκφραση αγαπητή στον πρόεδρο του Συμβουλίου η ιδέα είναι ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να οικοδομηθεί εις βάρος των κρατών μελών πόσο μάλλον εις βάρος των ιδίων των πολιτών γνωρίζετε κάποιον εσείς που θα μπορούσε να είναι αντίθετος με αυτή τη συνεργασία χωρίς φυσικά να διακινδυνεύσει διαψευστεί από τους εκλογείς του και να χάσει την νομιμότητα της ε, αντιπροσωπευσής του. Παρ' όλα αυτά η διαδικασία δεν είναι τέλεια, δυναμίες έχει, είναι αργή, είναι περίπλοκη και μερικές φορές και είναι πηγή θα έλεγα ε, πολλών προβλημάτων. Τα γνωρίζω πολύ καλά αυτά γιατί προέρχομαι από μια χώρα που απαιτεί την επικύρηση την επικύρωση μάλλον της συνθήκης από 7 διαφορετικά νομοθετικά σώματα. Παρ' όλα αυτά η διαδικασία αυτή έχει την δυνατότητα να ενημερώνει όλους τους υπεύθυνους πολιτικούς, να προκαλεί συζητήσεις με τους πολίτες της Ένωσης και να παρουσιάζει τις αποφάσεις στο κοινό της κάθε χώρας στα πλαίσια των ευρωπαϊκών πολιτικών η αμοιβαία εξάρτηση ανάμεσα από τη μία την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη τις εθνικές διοικήσεις πρέπει να είναι αποτελεσματική. Ο ατυπικός χαρακτήρας της ευρωπαϊκής για να επανέλθω σε αυτό που έλεγε ο Τελόρ είναι σαν διαστημόπλιο μη αναγνωρίσιμο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μας οδηγήσει στο να φανούμε πιο αυστηροί στις συγκριτικές μελέτες που κάνουμε για την κατάσταση των πραγμάτων. Μετά από τις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές και με το ποσοστό συμμετοχής να περιορίζεται στο 43% τέθηκαν πάρα πολλά ερωτήματα σχετικά με την προσμέτρηση αυτής της αυξανόμενης αδιαφορίας των ευρωπαϊκών πληθυσμών. Δεν θα επανέλθω στις διαφορετικές αιτίες τις οποίες γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Παρ' όλα αυτά η οικονομική κατάσταση είναι πολύ πιο ανησυχητική. Κανένας δεν έχει ξεχάσει τις διαδηλώσεις στην Ελλάδα σαν παράδειγμα. Όλα αυτά επηρεάζουν τις λήψεις αποφάσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξη ε, στη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και στα πλεονεκτήματα τα οποία προσδίδει στην κάθε χώρα μπαίνει μειούμενη. Νομίζω ότι η εμπιστοσύνη Σας ευχαριστώ πολύ για την ομιλία σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρόεδρε της Βουλής ε, του Βελγίου, θα ήθελα και πάλι να τονίσω, λέει ο πρόεδρος του σώματος, ότι έχουμε κοινή ευθύνη για το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο μετά από την επικύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας. Είναι μια ευθύνη την οποία αναγνωρίζουμε βεβαίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα έχετε τη δυνατότητα να συζητήσετε τις πτυχές της νομοθεσίας κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ε, του νομοθετικού έργου. Βασίζουμε λοιπόν στην συνεργασία σας ε, και κατά τη διάρκεια της σύνταξης των νομοθετικών πράξεων αλλά και κατά την περίοδο της εφαρμογής και υλοποίησης. Θέλουμε λοιπόν όλοι εμείς να υποφεληθούμε από την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ο κύριος Πρόεδρος είναι σήμερα μαζί μας για τη συζήτηση. Αύριο θα είναι και ο Πρωθυπουργός του Βελγίου μαζί μας, ο κύριος Ιβ Λετέρμ. Δεδομένου το Βέλγιο έχει και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο κύριος ε, Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εκτελεστικής Επιτροπής Κομισιόν. Το πρωί αύριο θα είναι παρόντες και επίσης ο, ο κύριος Πίτερς, ο πρόεδρος του Βελγικού, της Βελγικής Γερουσίας θα είναι παρόν. Επίσης θα ήθελα να προσθέσω ότι ε, έχουμε τρεις ομάδες εργασίες που θα συνεδριάσουν μετά από τη συζήτησή μας εδώ στην Ολομέλεια και θα ε, συνεδριάσουν οι ομάδες αυτές ξεχωριστά, αυτές οι τρεις ομάδες. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ζαν Πιέρ Ζουγέ, ο οποίος είναι πρόεδρος της αρχής εποπτείας ε, των ε, χρηματοπιστωτικών αγορών και επίσης στη Γαλλία και επίσης ήταν στη Γαλλία πρώην υπουργό ε, Εσωτερικών ε, ε, Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Πρόεδρε Μπουζέκ, κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων του Βελγίου, αγαπητέ Αντρέφλαο, Κύριε Ντεκρό, εκπρόσωπε της Βελγικής Προεδρίας που χαιρετίζω εδώ σήμερα, όπως και τον κύριο Φλό. Κυρίες και κύριοι βουλευτές από το Εθνικά Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αγαπητοί φίλοι Ευρωπαίοι, πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας. Πρέπει να σας πω ότι η παγκοσμιοποίηση που γνωρίζουμε σήμερα και που επηρεάζει ολόκληρη την Ευρώπη, το είπε και ο πρόεδρος Μπούζεκ και ο πρόεδρος Φλέο, μοιάζει πάρα πολύ με τη διεθνοποίηση που χαρακτήριζε τον πλανήτη μας στην αρχή του 20ου αιώνα. Στην αρχή, συγγνώμη, του, ναι, του 20ου αιώνα ο καθένας νιώθει ότι υπάρχει μια μεταφορά του κέντρου Βάρου, του πλούτου και της ισχύω μακριά από την Ευρώπη. Και ο λόγος δεν είναι ότι η Ευρώπη είναι πιο αδύναμη, αλλά ότι άλλοι φαίνονται περισσότερο ισχυροί. Αυτό συνέβη με αρκετέ από τις χώρες μας. Το ολικόφως του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου ήταν αυτό που έγινε με την Αγγλία και τη Γαλλία απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό που γίνεται σήμερα με την Ευρώπη απέναντι στην Κίνα, την Ινδία, τη Βραζιλία ή την Ρωσία. Βέβαια και οι Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν βαθμό αντιμετωπίζουν το ίδιο φαινόμενο. Η οικονομική κατάταξη των εθνών θα έχει ριζικά αλλάξει το 2020 και η αλλαγή αυτή υποχρεώνει την Ευρώπη να ανανεώσει τις σχέσεις της με τους μεγάλους της εταίρους. Και το κάνει. Το κάνει προσπαθώντας να βρει μια ισορροπία ανάμεσα σε μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση και την τάση, τον πειρασμό που έχουμε συχνά να σκεφτόμαστε ο καθένας για τον εαυτό του. Κάτι που είναι απόρρια βέβαια της ε, ισχύω του κράτους έθνους και σε ένα βαθμό και της διακυβερνητικής συνεργασίας. Η συνύπαρξη τώρα ενός ε, τρόπου κοινοτικής διαχείρισης και διακυβερνητικής βάζει πολλούς από τους εταίρους μας σε δύσκολη θέση. Χάνουν ε, λίγο πολύ τον μπούσουλα, δεν καταλαβαίνουν καλά πως έχουν τα πράγματα. Λείπει ο συντονισμός. Είναι περίπλοκες ιδέες. Τα και οι προηγούμενοι ότι η ανάγκη για Ευρώπη γίνεται περισσότερο αισθητή εκτός Ευρώπης παρά εντό Ευρώπη, γιατί ήδη οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Όλοι οι μεγάλοι θέλουν να έχουν ω εταίρο την Ευρώπη και θέλουν μια Ευρώπη που να βρίσκεται μέσα σε συγκεκριμένες δομές με τάξη και οι Ευρωπαίοι να μην μπαίνουν στον πειρασμό να ακούνε τις λαϊκίστικες ε, σιρήνες. Βρισκόμαστε μέσα σε κρίση, σε δημοσιονομική κρίση, σε κρίση του ευρώ και μέσα σε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο. Η Ευρώπη κατάφερε να σταθεί στο ύψο της, κατάφερε να διατηρήσει την επιρροή της. Τι προκλήσεις μένουν ακόμα για την Ευρώπη αν θέλει να πείσει πρώτα απ' όλα τους Ευρωπαίους πολίτες και στη συνέχεια τον υπόλοιπο κόσμο για αυτό ε, το οποίο κάνει. Άρα η Ευρώπη ποτέ δεν ήταν περισσότερο αναγκαία από ό,τι σήμερα. Είμαι πεπισμένο ότι η Ευρώπη δεν έχει να ντρέπεται για τίποτα. Έχουμε προκλήσεις μπροστά μας και η πρώτη πρόκληση που έχουμε είναι να πείσουμε τους εαυτούς μας ότι μπορούμε. Τότε θα πείσουμε και τους άλλους. Αποφύγαμε ένα σενάριο καταστροφής όπως είχαμε το 1929 και αυτό προσπαθώντας να αποφεληθούμε από ένα πλαίσιο συνεργασίας που έχουμε μεταξύ μας και από μια κοινή ευρωπαϊκή δράση. Ε, μην ξεχνάτε τι έγινε, τι έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία απέφυγε να βρεθούμε στην ίδια κατάσταση όταν πτώχευσε η Lehman Brothers. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επίσης με τόλμη αντιμετώπισε τις προκλήσεις και φρόντισε να βοηθήσει με ρευστό πολύ γρήγορα. Επίσης, ταυτόχρονα ενίσχυσε και τη συνεργασία της με όλες τις μεγάλες τράπεζες και μοίρασε στην Ευρώπη αμερικανικά δολάρια αλλά και αντίστροφα. Έτσι η Ευρώπη απέφυγε μια κατάσταση αλλά Lehman και έδειξε στον υπόλοιπο κόσμο ότι είναι σε θέση να αντιδράσει γρήγορα και με αποφασιστικότητα. Όσον αφορά τώρα την πραγματική οικονομία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα θυμόσαστε ότι έθεσε σαν ε, στόχο μια ανάκαμψη 1,5% του ευρωπαϊκού ΕΠ και τον πέτυχε το στόχο, τον ξεπέρασε μάλιστα, χωρίς ε, η διαφοροποίηση των μέσων που χρησιμοποιήθηκε να πλήξουν τις εθνικές οικονομίες ή την ακαιρότητα της εσωτερικής αγοράς. Έπειτα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, επιβλήθηκε σαν ένας κύριος εταίρος Ξάνοντα κατά 30 δισεκατομμύρια ευρώ τον όγκο των δανείων 2009-2010 για να στηρίξει την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και τι μικρέ και μεσαίες επιχειρήσει. Επίση, βοήθησε και η αλληλεγγύη μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Ε, θα θυμόσαστε τη στήριξη στη σωζήγια πληρωμών μελών ε, εκτός ευρωζώνης που πήγε από 12 στα 25 δισεκατομμύρια ευρώ και μετά από 25 σε 50 δισεκατομμύρια ευρώ και βοήθησαν επίσης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο μας επέτρεψε να δράσουμε με αλληλεγγύη και να σταθεροποιήσουμε τις χώρες που πλήγησαν περισσότερο από αυτή την κρίση. Επίσης η Ευρώπη επέβαλε και την μέθοδο του G20 και την ε, ατζέντα της μεταρρύθμισης έδωσε την προτεραιότητα καταρχήν στην καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων και στη μεταρρύθμιση του συστήματος ρυθμίσεων και εποπτείας και στην ενίσχυση του ρόλου των διεθνών δημοσιονομικών θεσμών. Η φωνή της Ευρώπης βάρινε στο G20 της Ουάσιγκτον και στο Λονδίνο στη συνέχεια τον Απρίλιο του 2009 και συνεχίζει να έχει μεγάλο βάρος και στη Σεούλ όπου καταφέραμε να πετύχουμε συμφωνία για μεταρρυθμίσεις με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, φροντίζοντα να υπάρχει μια νέα ισορροπία και να ανταποκριθούμε στην πραγματικότητα όσον αφορά το σχεδιασμό δυνάμεων. Η Ευρώπη νομίζω ότι κατάλαβε ότι για να αναλάβει τις ευθύνε της μέσα σε αυτή τη μεταρρύθμιση του παγκόσμιου καπιταλισμού έπρεπε να οργανωθεί και έπρεπε να οργανωθεί ώστε οι εταίροι της να ακούνε μία φωνή από την Ευρώπη. Και αυτό το υπογράμμισε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ευρώπη μπόρεσε να φτιάξει μια νέα αρχιτεκτονική της χρηματοπιστωτικής ρύθμισης με προληπτική εποπτεία για να ανταποκριθεί στην κρίση και να αποφύγει νέους συστημικούς κινδύνους. Αυτό είναι ένα όπλο, η αρχιτεκτονική αυτή, ένα όπλο που διαθέτει η Ευρώπη αναγκαίο στο διάλογο που έχει με τρίτες χώρες μέλη το G20. Η προληπτική υποπτία με τη δημιουργία των ε, τριών ε, οργάνων για τις τράπεζες, για τις ασφάλειες και για τις χρηματοπιστωτικές αγορές θα επιτρέψει την σωστή ευρωπαϊκή εποπτεία αρκεί να έχουν τα μέσα που χρειάζονται στη διάθεσή τους και την στήριξη και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων τώρα που ξεκινούν η δημιουργία τους. Πιστεύω ότι μπορέσαμε έτσι να αντιμετωπίσουμε μια δυσκολία που είχε η Ευρώπη για την οικονομική της ε, ολοκλήρωση. Η ρύθμιση των αγορών δηλαδή. Ήταν κάτι το οποίο δεν υπήρχε αρκετά στην Ευρώπη μέχρι τώρα. Άρα έχουμε τεράστιες ελπίδες με τη νέα αυτή αρχιτεκτονική ρύθμιση των ε, ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών. Το είπε και ο πρόεδρος εξάλλου νωρίτερα όσον αφορά την ατζέντα της Κομισιόν και τους στόχους των G20 για τα χρηματοπιστωτικά παράγωγα, για τους κανόνες της προληπτικής ρύθμισης, για τους οργανισμούς πιστοληπτικής ικανότητας, αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας κλπ. Τέλος, η Ευρώπη πρέπει να ξέρουμε ότι πετυχαίνει, παρά τις αβεβαιότητες που παραμένουν, Καταφέρνει όμως να αντιμετωπίσει και την κρίση των χρεών των κρατών μελών. Είναι αλήθεια ότι στην αρχή αντίδραση των 27 ήταν ε, αργή σε σχέση με το ρυθμό με τον οποίο προχωρούσαν οι αγορές. Τελικά όμως η Ευρώπη κατάφερε και την Ευρώπη την κατάλαβαν οι αγορέ. Το ευρώ σήμερα βρίσκεται στην ε, καλύτερη κατάσταση από ότι του τελευταίου πέντε μήνε. Δεν υπάρχει πια τόσο μεγάλη επιφυλακτικότητα από τι αγορέ και σε ένα μεγάλο βαθμό και η επιφύλαξη των επενδυτών σε σχέση με την Ελλάδα έχει έρθει. Όπω έχουν όμω τα πράγματα, η κρίση παραμένει. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η υπάρχει αδυναμία στην οικονομική διακυβέρνηση. Το είδαμε αυτό. Και αυτά προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε για να αποφύγουμε νέους συστημικού κινδύνους. Δεν υπήρχε πραγματικός μηχανισμός αλληλεγγύης για να βοηθάμε τις χώρες οι οποίες κινδυνεύουν με πτώχευση. Ε, απαγορεύαμε την διάσωση, τον bailout. Όμως με την απόφαση της 9 2010 για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Δημοσιονομικής Σταθερότητας φροντίζουμε να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα και ε, στη συνέχεια η Επιτροπή και ο κ. Φονροπάου πήραν εντολή να κάνουν προτάσεις προκειμένου να υπάρξει ένας μόνιμος μηχανισμός πια επίλυσης των κρίσεων πριν λήξουν τα προσωρινά μέτρα, ο προσωρινός μηχανισμός που λήγει το 2013. Προκειμένου όμως η απόφαση αυτή του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να γίνει πραγματικότητα, πρέπει να πάμε γρήγορα. Διότι ο χρόνο τη Ευρώπη, ο χρόνο δηλαδή που χρειαζόμαστε για να προσαρμόσουμε τι συνθήκε, δεν είναι ο ίδιο με τον ρυθμό τον οποίο προχωράνε οι αγορέ. Εξάλλου μπορεί να υπάρξουν και νέε πιέσει στα χρέη διαφόρων χωρών. Βλέπετε σήμερα τα ασφάλιστρα κινδύνου, τα επιτόκια, σε τι κατάσταση βρίσκονται και πόσο κινδυνεύουν οι περισσότερο ευάλωτοι παρά τα μέτρα λιτότητα που έχουν υιοθετήσει. Πρέπει επίσης να δώσουμε απαντήσει και σε δύσκολες ερωτήσεις. Τι μορφή πρέπει να έχει ο νέος μηχανισμός ε, για να αντιμετωπιστούν οι επίγουσες ε, ανάγκες που προκύπτουν. Ε, σε ποιες περιπτώσεις θα χρησιμοποιείται ένας τέτοιος μηχανισμός. Και τι θα κάνουμε με τις περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος πτώχευσης, πώς να αποφύγουμε οι αγορές ε, να μην πιέζουν ακόμα περισσότερο τις χώρες που είναι ευάλωτες. Και υπάρχει βέβαια πάβαλτα και το θέμα του ιδιωτικού τομέα. Πώς να αποφύγουμε επίσης την προπτική μιας ε, αυτόματης ε, βοήθειας να μην οδηγήσει άλλες χώρες να ακολουθήσουν διαφορετικές πολιτικές. Είναι πολύ λεπτά ζητήματα αυτά για τα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει φυσικά ένα λόγο μέσω της διαδικασίας συναπόφασης. Και νομίζω εδώ ότι η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι αποφασιστική σημασία για τις επόμενες συζητήσεις που θα έχουμε. Και υπάρχει και κάτι που μου φαίνεται ξεκάθαρο, είναι ότι δεν μπορούμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη στο σύστημα οργανωσή μα, στο σύστημα ρύθμισή μα, αν δεν φροντίσουμε να εφαρμόσουμε τον μηχανισμό αυτό δημοσιονομικών διευκολύσεων και αν δεν προβλέψουμε και αλλαγές της απλής δομής που είχαμε μέχρι τώρα σε άλλες θεσμικές ε, ρυθμίσεις. Βέβαια, δεν πρέπει να ντρεπόμαστε για τον απολογισμό που έχουμε μέχρι τώρα, καθ' άλλο. Πρέπει να ξέρουμε ότι ήμασταν 27 χώρες που καταφέραμε να συμφωνήσουμε για να πετύχουμε το αποτέλεσμα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι κανένας άλλος χώρος γεωγραφικά δεν έχει καταφέρει να επιδείξει ένα τέτοιο πνεύμα αλληλεγγύης και μια τέτοια ε, αντίδραση σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι πρέπει να επαναποφθούμε στις δάφνες μας. Προφανώς όχι. Όπως έλεγε και ο Ζακ Ντελόρ, η Ευρώπη είναι σαν ένα ποδήλατο. Αν ο ποδηλάτης ε, σταματήσει να γυρνάει τα πέταλια, πέφτει. Πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν, αλλά θα πρέπει να είμαστε και ξεκάθαροι ως προς τη ρότα που θα ακολουθήσουμε. Τι αυτή η περιπτώση θα πρέπει να αλλάξουμε και ταχύτητα ενδεχομένως, γιατί αλλιώς θα χάσουμε την επιρροή που έχουμε και θα χάσουμε και την υποστήριξη των πολιτών, όπως είπε και ο πρόεδρος Φλαό, λόγω της έλλειψης ε, φιλοδοξίας από πλευράς μας. Ποιες είναι οι προκλήσεις στις οποίες πρέπει να αντεπεξέλθουμε. Ε, η πρώτη παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο Πούσε και από τον πρόεδρο Φλεό. Ε, άλλη πρόκληση είναι η αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής δράσης και πώς γίνεται αντιληπτή από την κοινή γνώμη. Ε, είναι, έχουμε οργανωθεί ε, αυτά που ζητούν οι πολίτες για την απασχόληση, την ασφάλεια, την ε, δραστη, οικονομικές δραστηριότητες, την προετοιμασία του μέλλοντος. Η οικονομική και η χρηματοπιστωτική κρίση κατέδειξε ότι οι πρώτες απαντήσεις αναχέτησης της οικονομικής επιβράδυνσης ήταν μάλλον εθνικές παρά ευρωπαϊκές. Ε, δηλαδή, ο τρόπος λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη θα πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσει ε, της ε, σύγχρονης ε, διακυβέρνησης. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τα οικονομικά διαρθρωτικά προβλήματα, τα υπερβολικά ελλείμματα ή και τα πλεονάσματα, την αλληλεγγύη, καθώς και την ομοιομορφία των κανόνων στα πλαίσια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Αυτό μας παραπέμπει στο εργοτάξιο της οικονομικής διακυβέρνησης. Ακόμη όμως δεν έχουμε δει πραγματικές προτάσεις αποτελεσματικού συντονισμού των μακροοικονομικών πολιτικών. Τίποτα δεν προβλέπεται από αυτού για τη φορολογία. Από στην έκθεση που ε, υπέβαλε η κυρία Μπερέ, ε, τίποτα δεν προβλέπεται για τη φορολογία, για τον συντονισμό άλλων διαρθρωτικών πολιτικών, ούτε και των μέσων που θα επιτρέψουν στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν πολιτικέ που όμω δεν κατατείνουν προ τη συνεργασία με τα λοιπά κράτη-μέλη. Θα πρέπει να ρωτηθούμε για τι κοινωνικέ ευθύνε που καλούμαστε να υπομισθούμε, διότι λόγω τη κρίση έχουμε το θέμα τη ανακατανομή σε καλύτερο κατά μερισμού των προσπαθειών, ε, τη οριοθέτηση πολιτική μα στο επίπεδο κοινωνική προστασία, λειτουργία τη αγορά, ε, τη απασχόληση και τη χρηματοδότηση ε, των συντάξεων. Πέρα από τη διακυβέρνηση και το περιεχόμενο των πολιτικών που χαρακτηρίζει τη σχέση Ένωση με την κοινή γνώμη, όπω είπε και ο Πρόεδρο, βλέπουμε μια αποστασιοποίηση από πλευρά των πολιτών, την οποία υποτιμούμε. με την παγκοσμιοποίηση παγιώνεται η ανάγκη για την Ευρώπη, αλλά δεν υπάρχει επιθυμία για περισσότερη Ευρώπη Οπότε έχουμε και μία πρόκληση ως προς τους πολίτες, ε, δηλαδή ε, ε, η Ευρώπη αναλαμβάνει όλα και περισσότερες ευθύνε στην καθημερινή ζωή, παρόλα αυτά δεν θεωρούν ότι έχει οργανωθεί επαρκώς η Ελλάδα για, νέα, για να εξυπηρετήσει αυτή τη νέα ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Θα πρέπει βράχει πρόθεσμα λοιπόν να προβλέψουμε ώστε να τροποποιηθεί σχετικά η συνθήκη με την απλουστευμένη διαδικασία. Δεύτερη πρόκληση αυτή της χρηματοδότησης. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα του Κοινοβουλίου και τα εθνικά κοινοβούλια διαπιστώνουν ότι υποχωρεί ο ε, προϋπολογισμός της Ένωσης ε, και Κάποιοι ε, ε, το καταλογίζουν στους ευρωπαϊκούς ηθήνοντες, ε, στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι δεν έχει τα απαιτούμενα μέσα. Τώρα, εάν έχουμε ευρωπαϊκούς κανόνες, αλλά δεν έχουμε τα απαιτούμενα μέσα, ούτως ώστε με άμεσο και ορατό τρόπο να δρούμε αμελητή, θα χρειαστεί να καταβάλουμε μια επιπλέον προσπάθεια ως προς τον προϋπολογισμό της Ένωσης, μειώνοντας εδραστικά τα ελλείμματα, διότι και επενδυτές περιμένουν σαφή σημάδια σχετικά με τις προσπάθειες που θα γίνουν για τη μείωση των ελλημάτων. Δεν είναι απλή η απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι με ορθολογικό τρόπο πρέπει να αντιληφθούμε τη σημασία του ζητήματος και να καλύψουμε τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο επίπεδο ολοκλήρωσης ε, της Ευρώπης ε, και το χάσμα λοιπόν με τα μέσα που χρειαζόμαστε για να υλοποιήσουμε τις δράσεις που οφείλουμε να αναλάβουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν αποτιμώ καθόλου την ε, δυσκολία αυτής της πρόκλησης. Ε, κατόπιν, οι σχέσεις ανάμεσα στην Ευρώπη και στις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες. Δεν έχουμε οργανωθεί, δεν έχουμε συνταχθεί επαρκώς, ενώ ανοίγει η προοπτική ενός G2, ε, G4, δεν είναι κάτι εξωπραγματικό αυτό. Βλέπουμε τι γίνεται στις οικονομικές σχέσεις Κίνας-ΥΠΑ ε, στο εμπορικό μέτωπο οξύνονται οι αντιπαραθέσεις ε, και ε, ενισχύει οι διμερείς και όχι πολυμερείς σχέσεις. Η Ντόχα χαρακτηρίστηκε από αυτήν την ανεφροηγουμένου αύξηση της δύναμης των οδειόμενων οικονομιών ε, και της ανεφροηγουμένου οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η κοινή προσέγγιση είναι αδύνατη διότι δεν υπάρχουν εμπορικές αντιπαραθέσεις και οι επιπτώσεις που έχουν ως προ την απασχόληση. Υπήρχε στην αρχή μια συνολική η οποία όμως υποχώρησε λόγω των διαφορετικών οικονομικών κύκλων και της εξάρτησής μας από τις εξαγωγές και από το ε, επίπεδο ανάπτυξης ε, των οικονομιών μας. Ε, εμφανίζονται προστατευτικές τάσεις στον χρηματοπιστικό, γεωργικό και ενεργειακό τομέα στην Ευρώπη. Τέταρτη και τελευταία πρόκληση. Πώς μπορούμε να έχουμε τα ίδια αναπτυξιακά περιθώρια που θα μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε θέση απασχόλησης και πώς οι αγορές μπορούν να εξυπηρετήσουν την πραγματική οικονομία. Ε, γιατί αυτό είναι ο λόγο ύπαρξη ε, των αγορών, να χρηματοδοτούν τι πραγματικέ οικονομικέ ε, δραστηριότητε. Όμω οι ιδιώτε και τα θεσμικά όργανα έχουν κουραστεί από την αδιαφάνεια και από τη μεταβλητότητα των αγορών και Βλέπουμε τι γίνεται με τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου στη ΣΥΠΑ, με τα αξιόγραφα των κρατικών χρεών στην Ευρώπη. Προσπαθήσαμε να τα διαφοροποιήσουμε, να μην έχουμε μόνο κρατικό δανεισμό, αλλά πρέπει να βρούμε και αγοραστέ. Επίση, οι μεταβλητέ που υπήρχε στην αγορά των μετοχών, δυστυχώ μπορεί να μετακυλιστεί και στι αγορέ των ομολόγων. Ε, αποταμίευση, η οποία όμω δεν επενδύεται στην έρευνα και στην ανάπτυξη, στι μακροπρόθεσμε επενδύσει, στη μετα ε, ε, των ε, ε, βιομηχανιών μας που δυστυχώς καταναλώνουν υπερβολική ενέργεια. Ο πρόεδρος πλέον το τόνισε. Για να έχουν εμπιστοσύνη οι αγορές θα πρέπει ε, άρδιν να αναθεωρήσουμε την οδηγία για, τις, για τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τις αγορές που καλύπτουν και να διορθώσουμε παίρνοντα κάποιε αποστάσει ε, τι πλέον βλαβερέ συνέπειέ του. Σε παραδείγματο χάρη κατακαιρματισμό τη ρευστότητα και αυξανόμενη αδιαφάνεια των συναλλαγών ε, που επηρέασαν ακόμη και τα dark pools, τα υπονομαζόμενα, τι αδιαφανεί πηγέ ρευστότητα. Ε, υπάρχουν πιθανά διαρθρωτικά μέτρα για, μέσω τη προδιαπραγμάτευση Φερρυπίν να ανακοινώσουμε τι πρόκειται να κάνουμε, αν θα αγοράσουμε ή θα πουλήσουμε και με τα μέτρα μετά τη διαπραγμάτευση, μετά τη συναλλαγή. Δηλαδή τι αγοράζαμε, τι πουλήσαμε, ε, ποιο όγκο αξιογράφων, για ποια αξία. Επίση έχουμε τι τεχνολογικέ προκλήσει, τι αίσθηση λειτουργία των αγορών, δεδομένε και τη ανάπτυξη των συναλλαγών που υλοποιούνται από του high frequency ε, συναλλασσόμενου ε, στα χρηματιστήρια, με πολλέ συναλλαγέ δηλαδή. Υπάρχουν πάρα πολλέ τέτοιε τεχνικέ που συνεπάγονται κινητοποίηση επενδύσεων και κεφαλαίων ιδιαίτερα υψηλών, ε, αλλά η κοινωνική τους ωφελημότητα μπορεί να αφασβητηθεί ε, δεν θα πρέπει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να φοβάται ε, τις ε, φιλοδοξίες που πρέπει να έχουμε σε αυτούς τους τομείς. Επίσης ε, να είμαστε φιλόδοξοι για την οργάνωση των νέων αγορών. Όπως αυτά που συμβαίνουν στις ΗΠΑ έτσι και στην Ευρώπη μπορούμε να επηρεάσουμε τις εργασίες του G20 που ευτυχώς ε, ή δυστυχώς θα πρέπει να επιληφθεί του ζητήματος, αλλά είναι σαφές ότι η υποδειγματικότητα του ρόλου της Ευρώπης θα είναι συνάρτηση των φιλοδοξιών που θα έχει για την αναθεώρηση αυτής της οδηγίας για τις αγορές του χρηματοδοτικού μέσου. Ας μην ξεχνάμε επίσης την οργάνωση των νέων αγορών. Αύριο θα έχουμε αγορές του διοξιδίου του άνθρακα, των ενεργειακών παραγόγων, ε, διατροφικών παραγόγων που όλο ένα και παγκοσμιοποιούνται και είναι λυπής η εποπτεία τους προς το παρόν και οι κερδοσκοπικές μεθοδεύσεις αναφέρονται σε αυτές τις αγορές ε, συχνά. Ε, η Γαλλία έχει αναλάβει την προεδρία του G20 και θα επιληθεί αυτού του ζητήματος της ρύθμισης των αγορών που έχουμε παραμελήσει μέχρι τούδε. Ε, βλέπουμε εδώ και πάλι ότι είναι εκ των όνου η οργάνωση, είναι μάλλον αδύρυτη ανάγκη η οργάνωση αυτών των αγορών. Να ξαναβρούμε λοιπόν την ανάπτυξη που είχαμε στο παρελθόν και από αυτήν την ε, πλευρά πολλές προτάσεις ε, του Επιτρόπου Μπαρνιέ έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, ιδιαίτερη σημασία. Ε, υπάρχουν δε πολυάριθμες συστάσεις από εργασίες που έλαβαν χώρα πριν από χρόνια σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα ε, για την ε, πολιτική για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή ε, για την πολιτική προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων παραδείγματο χάρη διότι ο πλούτος μας είναι λικός και άειλος περισσότερο από το παρελθόν και εμεί σας πω περισσότερο άειλος οπότε έτσι μπορούμε να καινοτομήσουμε, να δημιουργήσουμε νέες ιδέες, νέα εργαλεία για να έχουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα έχει καταλητικό ρόλο για τις αναπτυγμένες οικονομίες. Ταχύτατα πρέπει να παίξουμε αυτό το χαρτί, να άρουμε τους φραγμούς όταν υπάρχουν και να δημιουργήσουμε τα επιτούτο εργαλεία όταν δεν υπάρχουν για να υλοποιήσουμε αυτές τις πολιτικές. Τέλος, ένα από τα 50 μέτρα που προβλέπονται σε αυτό το σύμφωνο των ενιαίων αγορών είναι αυτό που αποσκοπεί στην πρόσβαση της, ε, τη βελτίωση μάλλον της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στι αγορές. Ε, κατά προτεραιότητα θα πρέπει να μέσα από το Small Business Act οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τις ε, αγορές ε, όπως είχε προταθεί και από την κυρία Λαγκάρ και από τον κύριο Σόμπλε Σόιμπλε ε, και όλα αυτά προφανώς θα πρέπει να χαρακτηριστούν από διαφάνεια και να τονίσουμε και την ανάγκη που υπάρχει να λαμβάνουμε υπόψη την οπτική γωνία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, για να καλύψουμε αυτές τις ε, απαιτήσει που υπάρχουν για την εποπτεία και να τις προσαρμόσουμε στο μέγεθος αυτών των επιχειρήσεων. Ιδού κάποιες από τις προκλήσεις ε, που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει τους επόμενους μήνες και χρόνια η Ευρώπη. Σας μίλησα για το πάγιο ερώτημα του ρόλου του ευρώ που βρίσκεται σε πολύ υψηλά ή σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ε, επίσης, ε, αμυντική βιομηχανία, το πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη, ποια είναι τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρώπης, πώς θα υπεραμεινθούμε αυτών των συμφερόντων, πώς θα ε, έχουμε πιο εξορθολογική διαχείριση του, του ομέα αυτού, που δεν είναι ο μόνος. Υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς για τους οποίους οι εταίροι μας μας ζητούν περισσότερη σαφήνεια, περισσότερη συνέπεια. Πρέπει λοιπόν να αποδείξουμε ότι μπορούμε να οργανωθούμε και θα κρυθούμε από τα αποτελέσματα των δράσεών μας, από το ε, μέτρο στο οποίο θα μπορέσουμε να προσαρμοστούμε σε ένα νέο διεθνές ε, περιβάλλον, οικονομικό περιβάλλον, αμυντικό περιβάλλον, γιατί εξαρτώμαστε από τον υπόλοιπο κόσμο. Η Ευρώπη θα πρέπει να υπερβεί, ε, να κάνει υπερβάσεις και όχι να υποχωρήσει και να συνάγω ότι η ουτοπία τελικά μας οδήγησε σε μια υποχώρηση, ε, οδήγησε την Ευρώπη στο να σηκώσει τα χέρια ψηλά. Ε, δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε μπροστά σε αυτόν τον ε, νέο φιλελευθερισμό της Ευρώπης. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η σημερινή συζήτηση ταιριάζει, είναι πάρα πολύ κατάλληλη με όλες τις άλλες συνεδριάσεις που γίνονται εκ παραλίλου στην Ευρώπη για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Εκ των υστέρων βλέπουμε πόσες λεπτομέρειες χρειάστηκαν για να διαμορφώσουμε τις συζητήσεις μας και σε πόσες λεπτομερείς πτυχές πρέπει να, να μπούμε, πρέπει να εισέλθουμε όπως θα δείτε στις τρεις ομάδες εργασίας για να διατυπώσουμε τις απαντήσεις. Όπως είπε και ο πρόεδρος κύριος Μπούζεκ, χρειαζόμαστε δράση, χρειαζόμαστε να ενεργοποιηθούμε, να δράσουμε πάρα πολλές αποφάσεις θα ληφθούν σε εθνικό επίπεδο και θα είναι αποτελεσματικές. Αυτό είναι σίγουρο. Έχουμε όμως και χρονική πίεση, οπότε ορισμένα σημαντικά θέματα θα τα περάσουμε μόνο στο γόνατο σήμερα. Άρα λοιπόν έχει μεγάλη σημασία να κάνουμε συζητήσεις σε βάθος. Συζητήσεις με στοιχεία, συζητήσεις ε, ενδελεχείς οι οποίες θα μας δώσουν τη δυνατότητα με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Ε, υπάρχουν χώρες που βρίσκονται ας πούμε στην ανάκαμψη αλλά υπάρχουν άλλες χώρες που αυτή τη στιγμή πονάνε ή βρίσκονται μέσα στο επίκεντρο της κρίσης. Άρα λοιπόν οι ενέργειες που πρέπει να κάνουμε για την ολοκλήρωση της εσωτερικής, της κοινή αγοράς και για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής του 2020 θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους περιορισμούς του προϋπολογισμού και τους, του, τις, τους περιορισμούς, της περικοπές που πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δημόσιες ε, περικοπές ε, ελπίζω να μην οδηγήσουν στην ακύρωση ή κατάργηση πάρα πολύ σημαντικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος θέτουμε πάντοτε φιλόδοξους και υψηλούς στόχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραδείγματο χάρη, οικονομική ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας και άλλους. Όμως μας λείπει το όραμα, το μακροπρόθεσμο και παγκόσμιο. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πιστεύω ότι το πρόγραμμα Ίντερ θα μπορέσει να καλύψει το χάσμα, το κενό μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και, και της υπόλοιπης υφηλίου. Πιστεύω ότι ο καινούργιος προϋπολογισμός για τη νέα ε, και οι νέες δημοσιονομικές ε, προοπτικές θα μπορέσουν να παράσχουν αυτήν τη μακροπρόθεσμη παγκοσμιοποιημένη προοπτική. Πώς θα επιτύχουμε λοιπόν αυτές τις μεσοπρόθεσμες παραμέτρους ε, για να ολοκληρώσουμε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 2020. Παραδείγματος χάρη το 3% του ΑΕΠ ε, να διατεθεί σε στις επιστήμες και στην έρευνα και να μην το περικόψουμε. Ευχαριστώ. Μιλήσατε ταχύτατα και έτσι σεβαστήκατε το χρόνο ομιλία σας, λέει ο Πρόεδρος. Υπάρχει ε, μια μπλε κάρτα, κάποιος με μπλε κάρτα. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Λίνο Βίλιο από την Ιταλική, μέλος της Ιταλικής Βουλής. Βουλής. Πράγματι η οικονομική κρίση μας έχει επιβάλει σε όλους την ανάγκη να συνεχίσουμε την προσπάθεια της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης. Αντίθετα από τα τελευταία περιφατικό θα έλεγα πρόγραμμα των συνταγματικών ρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ τώρα έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις να κάνουμε πραγματικότητα τις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών να κάνουμε πραγματικότητα αυτά που έλεγε ο Ζωάν Μονέ ότι μόνο η οικονομική συνεργασία με μια συγκεκριμένη μορφή αλληλεγγύης ανάμεσα στις διάφορες χώρες θα μπορέσει να αποδείξει ότι η Ευρώπη είναι απαραίτητη. Γι' αυτό και η στρατηγική του 2020, η οικονομική διακυβέρνηση και η εσωτερική αγορά μπορούν να μας βοηθήσουν να πετύχουμε τον συγκεκριμένο στόχο. αρκεί τα ευρωπαϊκά όργανα και τα εθνικά όργανα να έχουν το θάρρος το οποίο μέχρι τώρα ίσως δεν είχαν όλοι. πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με την οικονομική κρίση και να μην κολλήσουμε στο τοτέμ θα έλεγα της σταθερότητας. Δεν θα πρέπει να μιλάμε μόνο για τα ανώτατα όρια οικονομικής παρέμβασης αλλά για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών των οικονομικών παρεμβάσεων. Συμφωνώ επίσης με αυτούς οι οποίοι είπαν ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στον τομέα των φορολογικών ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη. Συμφωνώ με την ιδέα του κατωτάτου φορολογικού ορίου, σαν παράδειγμα, ποσοστού. Μου φαίνεται επίσης ότι υπάρχουν ελλείψεις στη στρατηγική του 2020 για την ε, οικονομική governance απουσία προτάσεων για την ενιαία παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Νομίζω βέβαια Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφοι. Δεν βλέπω μπλε κάρτα, οπότε συνεχίζω και δίνω το λόγο στην κυρία Ντάνα Φαχάλοβα. Α, μπλε κάρτα. Παρακαλώ, πείτε ποιο είστε όμως πρώτα. Εγώ σας ξέρω, αλλά πείτε ποιο είστε παρόλα αυτά. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Βίλεφ Τσέφτερ, πρόεδρο τη Επιτροπή Βαγκοπιθέσεων ε, του Τσεχικού Κοινοβουλίου. Θα συνεχίσω στα τσεχικά, αν μου επιτρέπετε. Θέλω να ευχαριστήσω τον προλαλήσαντα. Αλλά θέλω να ρωτήσω, τι το κακό είναι οι φόροι. Μιλάμε για χαμηλούς φόρους, αλλά τότε δεν έχουμε έσοδα με, από τους φόρους. Απαντήστε παρακαλώ. Εγώ μιλάω για τον ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών στο φορολογικό επίπεδο. Πρέπει να προβλέψουμε ένα ελάχιστο επίπεδο φορολόγησης ώστε να αποφύγουμε χώρες εξαιτία της εσωτερική τους κατάστασης να επιβάλλουν ε, φορολογικούς συντελεστές ε, που να είναι τέτοιοι που να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν δεν υπάρχει ρύθμιση θα υπάρχει ένας αγώνας δρόμου μεταξύ των χωρών μελών σε βάρος των πιο φτωχών. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρχει αν όχι η ομοιομορφία, τουλάχιστον ένα συντονισμό τη φορολογική πολιτική. Συμφωνώ με αυτά που υπόθηκαν πριν, ότι πρέπει να σκεφτούμε μήπω έχουμε έναν ελάχιστο συντελεστή κάτω από τον οποίο να μην κατεβαίνουμε για να αποφεύγουμε ακριβώ τέτοιου είδου ε, αθέμητο ανταγωνισμό. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Τώρα η κυρία Ντάνα Βαχάλοβα έχει το λόγο παρακαλώ. Από το Κοινοβούλιο της Τσεχίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, ζούμε σε μια εποχή όπου η παγκόσμια οικονομία έχει χτυπηθεί από την οικονομική κρίση. Βλέπουμε τράπεζες να καταραίουν, επιχειρήσεις να καταραίουν και το ερώτημα είναι πώς διαδεχειριστούμε αποτελεσματικά την κρίση. Κανένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να το επιτύχει αυτό από μόνο του. Αλλά η αηφόρος ανάπτυξη την οποία επιδιώκουμε δεν μπορεί να βασιστεί σε βραχυπρόθεσμες λύσεις και να είναι μόνο οικονομικές αυτές οι λύσεις ε, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι η κερδοφορία είναι ο βασικός στόχος ε, του επιχειρηματικού κόσμου. Και αυτό δεν εγγυάται την ευημερία των πολιτών μας. Η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται στην επίτευξη αηφόρου ανάπτυξης. Και όταν λέμε αηφόρος ανάπτυξη εννοούμε ότι αυτό είναι το κλειδί της υγιούς ανάπτυξης. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει και νοοτροπία, να σπαστεί αυτή, αυτό το στόχο η Ευρωπαϊκή Ένωση, παραδείγματο χάρη τώρα που πολεμούμε όλοι για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήματος. Δεν είναι μόνο οικονομικά τα στοιχεία που επιδιώκουμε, πρέπει να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών, να εξασφαλίσουμε το μέλλον των, των επόμενων γενιών, των παιδιών μας και αυτοί οι οποίοι διαδίδουν το μήνυμα ότι κάθε θεραπεία της κρίσης βασίζεται μόνο στην ανάνυψη της αγοράς κάνουν λάθος. Είπαμε ότι κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί μόνο να αντιμετωπίσει την κρίση, αλλά η ανάπτυξη καινοτόμου και καινοτόμων κλάδων και επιχειρήσεων βοηθάει. Γι' αυτό η κινητήρια, εάν η κινητήρια δύναμη για το ΑΕΠ, για όλα τα ΑΕΠ, είναι η επίτευξη κερδών του επιχειρηματικού κόσμου δεν θα ξεπεράσουμε την κρίση. Ιδίω σε χώρες που έχουν ε, πληγωθεί πάρα πολύ στο, στην Ευρώπη βλέπετε ότι είναι χώρες που έχουν ε, αναπτύξει καλές υποδομές, καλές βιομηχανίες και όμως ένα καλό επιχειρηματικό κλίμα και όμως έχουν θυγεί πάρα πολύ. Άρα λοιπόν η συνεχής επιδίωξη ε, χρηματοοικονομικών στόχων δεν βοηθάει και αυτή την οτροπία πρέπει να σπαστούμε. Πρέπει να συντονίσουμε τα κοινωνικά μέτρα με τα οικονομικά, διότι η καλή ευρωπαϊκή διακυβέρνηση δεν είναι μόνο δημοσιονομική πρέπει εκ παραλίλου να βοηθήσουμε τους πολίτες μας να ε, αναπτύξουν μια υγιή κοινωνία και μια υγιή αγορά εργασίας. Ευχαριστώ. Ε, κάποιος έχει μπλε κάρτα. Ναι, είναι καλύτερα να σας δω άμα τη σηκώσετε και να, να δω ποιος είστε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο προηγούμενος ομιλητής ε, ανέφερε την ανάπτυξη ε, των επιχειρήσεων του επιχειρηματικού κόσμου που, η οποία θα πρέπει να βασίζεται στην αηφόρο ανάπτυξη και δεν υποστήριξε ιδιαίτερα την κερδοφορία ή μάλλον την επιδίωξη του κέρδους όμως, ε, μία υφόρος ανάπτυξη επιχειρηματική πρέπει να βασίζεται στο κέρδος. Πώς μπορούμε λοιπόν να ε, ε, υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις να επιδιώξουν και να επιτύχουν την αηφόρο ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ για να απαντήσετε κύριε Βαχαλόβα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε κίνητρα σε επιχειρήσεις με πολλούς τρόπους. Με πολλά σχέδια τα οποία τις κάνουν να δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης. Αυτό βέβαια πρέπει να γίνει και σε άλλο επίπεδο και σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόεδρο, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα ο φίλος μου Πιέρ Λεκιγέρε έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να πω ότι ο Ζων Πιέρ Ζουγέ έδειξε παραδειγματικά με ποιο τρόπο η Ευρώπη αντέδρασε θετικά στην κρίση. Έχουμε συχνά την τάση να επικρίνουμε την Ευρώπη. Ε, η Ευρώπη όμως τέσσερις φορές παρενέβη σε μεγάλες κρίσεις που όπως είπε και αυτός νωρίτερα θα μπορούσαν να μας είχαν ε, οδηγήσει στην κατάσταση του 1929. Όχι όμως, η Ευρώπη μπόρεσε να αντιδράσει. Δεύτερον, συμφωνώ επίσης για το ότι πραγματικά σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται όσο ποτέ. Πριν από τρία-τέσσερα χρόνια λέγαμε ο κόσμος αλλάζει, υπάρχουν εξελίξεις. Ε, λοιπόν σήμερα τις έχουμε τις εξελίξεις. Είναι μπροστά μας, τις βλέπουμε κάθε μέρα. Ε, βλέπουμε ε, να εμφανίζονται νέες ε, δυνάμεις, νέες χώρες. Γι' αυτό λέμε ότι η Ευρώπη χρειάζεται σήμερα όσο ποτέ. Ήταν πολύ θετικό το βήμα που έκανε στις 29 Οκτωβρίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που υιοθέτησε την ε, έκθεση της Task Force υπό τον πρόεδρο Φανουροπάη. Επίσης, έτσι μπορούμε να ανταποκριθούμε στο θέμα της ανταγωνιστικότητας χάρη στην συνέχιση του μηχανισμού με άλλο τρόπο διάσωσης. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η διακυβέρνηση. Εδώ θέλω να αναφερθώ στην έκθεση Καρέ Σερβιγιών που έκανε η Επιτροπή, της οποίας εγώ προεδρεύω, στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Και θέλω να επιμείνω επίσης για το ότι η Ευρώπη τελικά έχει βγει ενισχυμένη από το στάδιο αυτό. Το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου θα πρέπει να συμπληρώσει τις αποφάσεις. Όμως δύο παρατηρήσεις έχω να κάνω. Πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια μπορούν να βοηθήσουν ε, για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Τα Εθνικά Κοινοβούλια πρέπει να συζητούν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το εξάμεινο αυτό. Και γι' αυτό και ανέλαβα μια πρωτοβουλία με την Επιτροπή Οικονομικών της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης για να δούμε μήπως μπορούμε να προτείνουμε μια διακοινοβουλευτική συνάντηση ειδική κάθε χρόνο το Μάιο να γίνεται μια διάσκεψη για τον προπολογισμό όπου να συμμετέχουν οι υπεύθυνοι των Οικονομικών Επιτροπών των Εθνικών Κοινοβουλίων και ο πρόεδρος της Επιτροπής Προπολογισμών. Μια άλλη ιδέα επί της ουσίας τώρα. Πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να επενδύουμε αμοιβαία για το μέλλον όσον αφορά την έρευνα, τις ανώσιμες πηγές ενέργειας, την άμυνα. Νομίζω ότι θα πετύχουμε το στόχο μας μόνο εφόσον φροντίσουμε ο εθνικός προϋπολογισμός να είναι καλά συντονισμένος και να συζητήσουμε και το θέμα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει κάποιο σηκώσει πλέκαρτα. Θα δώσω την προεδρία στο φίλο μου την Κουέλμα και η καρέκλα Ευχαριστώ πολύ, Χέρμαν. Έχουμε διάφορους ομιλητές. Ο επόμενος θα είναι ο συνάδελφός μου, ο κύριος Ζαμπιέρ Οντί. Ευχαριστώ, κύριε ζητήσει να μην γίνονται τέτοιου είδου συνεδριάσει κατά τη διάρκεια τη εβδομάδα των πολιτικών ομάδων αλλά κατά τη διάρκεια τη εβδομάδα των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Και αυτό είναι πολύ περίπλοκο και πράγματι η παρουσία μας εδώ είναι σχετικά περιορισμένη θα έλεγα από πλευρά των συναδέλφων. Ο κύριος Πέτρου Φίλιπ τώρα από την Ρουμανική Γερουσία. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ όλους που βρισκόμαστε σήμερα εδώ μαζί για να συζητήσουμε το μέλλον της Ευρώπης, το οποίο είναι αναπόφευκτο, προς το μέλλον βαδίζουμε, είτε το θέλουμε είτε όχι. Και πρέπει να προβλέψουμε τι θα συμβεί μετά την κρίση το ερώτημα που θα μας θέσουν οι πολίτες μας είναι εάν μετά την κρίση θα έρθουν καλύτεροι καιροί. Θυμάμαι όταν ε, στην προηγούμενη εντολή του θητεία του Κοινοβουλίου ήμουν Ευρωβουλευτής επί Γαλλικής Προεδρίας στην Ολομέλεια του Στρασβούργου ο πρόεδρος Σαρκοζή είχε ανακοινώσει θριαμβευτικά την οικονομική κρίση στην Ευρώπη. Γύρω στις 15 Σεπτεμβρίου ήταν. Α, ναι, τρία λεπτά έχω να μιλήσω. Το, το βλέπω. Ε, αλλά όπως έλεγα, ο πρόεδρος Μπαρόσο είχε πει τότε λοιπόν, μετά από την επίσημη ανακοίνωση της κρίσης, είχε δημιουργήσει ο πρόεδρος της Κομισιόν μια ειδική επίτροπη που θα μελετούσε τις λύσεις ε, που πρέπει να εφαρμόσουμε για την αντιμετώπιση της κρίσης. Αναρωτιέμαι λοιπόν ε, αν αυτή η επιτροπή υπάρχει, αν υπάρχει, ε, αυτό είναι πολύ σωστό, πολύ καλό γεγονός, αλλά αν έχει βρει τις λύσεις και τις απαντήσεις. Η ουσία είναι ότι αυτή η συνάντησή μας, η συνεδρίασή μας σήμερα δεν πρέπει να είναι μία και μοναδική, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας στο μέλλον. Είτε μιλάμε για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε για τις ενέργειες των Εθνικών Κοινοβουλίων. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να οργανωθούμε όλοι μαζί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουμε να δώσουμε στους πολίτες μας να καταλάβουν τη λογική του νομοθετικού πλαισίου που ακολουθούμε. Για να καταλάβουν οι πολίτες μας ποια λογική διέπει το νομοθετικό μας έργο. Συγκεκριμένα ε, υπάρχουν ακόμα πολλοί φάκελοι που εκκρεμούν, οδηγίες που εκρεμούν, σε διάφορους τομείς όπως στην ενέργεια, στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, φάκελοι που αφορούν το Ταμείο Συνοχής, τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές 2013-2015, ε, και πολλοί άλλοι φάκελοι. Τώρα πάνω σε αυτούς του φακέλους έχει προσθεθεί και το βαρύτατο, φάκελο φάκελο φάκελος της οικονομικής κρίσης ε, που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Βεβαίω η Ρουμανία υποστηρίζει όλα αυτά τα πακέτα τα οποία τα τρία θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υποβάλουν προς είναι όμως πολύ σημαντική η συνέχιση αυτής της επικοινωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Η αξιοπιστία αυτών των φακέλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο διακυβεύεται. Υπάρχει ο κίνδυνος κατά τη διάρκεια μιας κρίσης οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που η πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο Ευχαριστώ. Βλέπετε, όταν παίρνετε εσείς το λόγο, μια που είσαστε βετεράνος εδώ, δεν μπαίνει μπρος το χρονόμετρο. Τώρα όμως το λόγο έχει ο Χάρη Φανμπόμελ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, Συμφωνώ με τον κύριο Φλό που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κάνει αρκετά για να στηρίξει, τη... να στηρίξει τα έσοδα και την ε, κατανομή τους την ισόρροπη. Διότι πολλά έκανε η Ευρώπη, αλλά δεν κατέληξε να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ανεργίας και να προστατεύσει τους ανέργους. Η πραγματικότητα στην Ευρώπη είναι, αλλά και στην Ολλανδία, είναι ότι οι κυβερνήσεις είναι έτοιμες να στηρίξουν τις τράπεζες, να στηρίξουν την αυτοκινητοβιομηχανία με χρήματα των φορολογούμενων, αλλά λίγα κάνουν για τους ίδιους τους πολίτες. Οπότε καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην Ευρώπη και φοβούμε ότι αν δεν αντιμετωπιστεί η ανεργία θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Έχω τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, δεν επήγει να γίνει μια αξιολόγηση της νεοφιλελεύθερης πολιτικής που εφαρμόζουμε στην Ευρώπη, την ελευθέρωση των αγορών που ονομάζεται και μετά την φιλελεύθερη πολιτική και η οποία έχει οδηγήσει στο να χάνονται χιλιάδες θέσεις απασχόλησης όπως γίνει στην Ολλανδία. Δεύτερον, δεν προβλέπουμε ότι ο σκεπτικισμός των πολιτών στην Ευρώπη θα αυξηθεί και ότι δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό αν δεν κάνουμε κάτι για τους ίδιους. Και τρίτον, εφόσον μειώνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Ευρώπη, δεν σημαίνει ότι και τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να βγάλουν το συμπέρασμα ότι υπάρχει λιγότερη αλληλεγγύη. Εγώ φοβάμαι ότι η κρίση στο δημοσιονομικό τομέα είναι λιγότερο σημαντική από την κρίση εμπιστοσύνης, η οποία θα οδηγήσει σε άσχημο δρόμο την Ευρωπαϊκή Ένωση που φτιάχτηκε για να μας οδηγήσει σε περισσότερη ελευθερία. Ευχαριστώ. Κλείνει εδώ ο κατάλογο των ομιλητών γιατί έχουμε πολλούς ακόμα, λέει ο Πρόεδρος. Και ακούσουμε και τον κύριο Ρουγέ. Παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο σας. Τρία λεπτά, όπως έκανε και ο τελευταίο ομιλητή. Τώρα, η κυρία Ολβίκη Λούνατσεκ έχει το λόγο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ως πρώην μέλος του Εθνικού Κοινοβουλίου χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω ορισμένου αυστριακούς συναδέλφους εδώ. Τώρα ως Ευρωβουλευτής θα ήθελα να επανέλθω σε ένα σημείο που αναφέρθη ήδη, α, ναι, στην έλλειψη παρουσιών ευρωβουλευτών εδώ, στην αίθουσα. Ήθελα να εξηγήσω ότι ε, ακόμα υπάρχουν επιτροπές που ασχολούνται με τα ίδια θέματα, ε, που όμως δεν συνεδριάζουν σήμερα, όπως η ΕΚΟΝ. Και αυτό ήθελα να διευκρινίσω και να πω ότι πραγματικά είναι γεγονός αυτό. Όσον αφορά τις ε, κοινέ συνεδριάσεις ε, Εθνικών Κοινοβουλίων με Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι λίαν χρήσιμες, ιδίω σε, σε περίοδους κρίσεων. Εμείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντοτε ζητούσαμε στενότερη συνεργασία στις οικονομικές πολιτικές και στενότερη εποπτεία παραδείγματος χάρη και εθνικών προϋπολογισμών πρέπει να εποπτεύουμε και να εξετάζουμε τα στοιχεία της Eurostar παραδείγματο χάρη. Έτσι, αυτός είναι ένας τρόπος να προλαμβάνουμε οικονομικές κρίσεις και γι' αυτό για να κάνουμε μια σωστή δημοσιονομική εποπτεία πρέπει να έχουμε τη βοήθεια των Εθνικών Κοινοβουλίων και των Εθνικών Αρχών. Παραδείγματο χάρη, ακόμα και οι διάφορε οικονομικέ επιτροπές ή υποεπιτροπές εθνικών κοινοβουλίων ή η Οικονομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να συνεργάζονται και να συνομιλεί με τις αντίστοιχες επιτροπές σε εθνικό επίπεδο. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει εθνική και ευρωπαϊκή συνεργασία στα διάφορα επίπεδα μεταξύ αρμοδίων επιτροπών το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προτείνει ισχυρότερες ε, προτάσεις, ισχυρές προτάσεις πρόβλεψης και ε, εποπτείας και ελέγχου των κρίσεων. Αλλά οι προτάσεις μας δεν έχουν ληφθεί υπόψη όσο θα έπρεπε. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ότι βλέπουμε την κρίση, την προοπτική της αντιμετώπισης της κρίσης με την ίδια οπτική γωνία. Ε, οι Βρυξέλλες όμως δεν έχουν καταφέρει να περάσουν αυτές τις ισχυρές ε, ιδέες που προτείναμε. Παραδείγματος χάρη το κείμενο των ε, ε, οικονομικών συναλλαγών, εποπτεία ε, οικονομικών συναλλαγών, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Δεν έχει περάσει ακόμα αυτή η πρόταση και πρέπει να πιέσουμε ισχυρότερα ε, και να επιτύχουμε καλύτερο συντονισμό. Αυτά τα, αυτές οι προτάσεις έχουν άμεση επίπτωση στην παρακολούθηση και εποπτεία του προϋπολογισμού και των εθνικών στοιχείων οι κυβερνήσεις υπό το νέο προϋπολογισμό χρειάζονται χρήματα ε, για να μπορέσουν να επενδύσουν περισσότερο στους τομείς της ενέργειας ε, για να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα και για να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Άρα λοιπόν οι εθνικές κυβερνήσεις χρειάζονται λεφτά, άρα πρέπει να έχουμε αυστηρότερο έλεγχο και εποπτείας ε, των πιστώσεων. Ευχαριστώ. Ο κύριος αλλά έχει σηκωθεί μία μπλε κάρτα. Κοιτάξτε, πρώτα θα ζητήσω από την κυρία τσεκ αν δέχεται την ε, ερώτηση. Την δέχεται. Λοιπόν, έχετε συνεπώς 30 λεπτά για να θέσετε την ερώτησή σας και 30 λεπτά για να δοθεί απάντηση. 30 δευτερόλεπτα, συγγνώμη, για να δοθεί είπατε ότι εφόσον υπάρξει μεγαλύτερος έλεγχος για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό τα πράγματα μπορεί να βελτιωθούν. Αυτό είναι κάτι το οποίο βέβαια μπορεί να αμφισβητηθεί διότι μπορεί να δημιουργηθούν περιπλοκές σε τομείς όπως η κατοικία, οι συντάξεις κτλ. Κοιτάξτε, για να λύσουμε την κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εσωτερική αγορά. Έχουμε ένα κοινό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλα αυτά υπάρχει ε, μια έλλειψη ελέγχου εθνικών προϋπολογισμών όπως αυτό συνέβη στην Ελλάδα και οι πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν για την κατάσταση των διαφόρων χωρών δεν είναι πάντα πλήρεις και έγκυρες. Δεν υπάρχει εδώ καμία πρόθεση παρέμβασης, αλλά θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με την κοινή της αγορά, με την ενιαία αγορά. Τότε θα πρέπει να υπάρξει σεβασμός των κανόνων. Ο Αλμπέρτο Κώστα από την Βουλή της Πορτογαλίας. Ευχαριστώ. Αυτή η ιδέα να χρησιμοποιήσουμε την κρίση και να προοδεύσουμε στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης είναι ευπρόσδεκτη. Είναι μια απαραίτητη ιδέα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποφύγουμε το εξή. Οι προϊούσες μεταρρυθμίσεις να πληγούν από ε, μηνύματα που δείχνουν ε, μία συμπεριφορά απρόβλεπτη. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα. Παραδείγματο χάρη, η αύξηση των ε, κυρώσεων. Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι πώς βλέπουν την διεύρυνση και την ε, αύξηση των ε, κυρώσεων θεωρούν ότι δίνεται μια αυστηρή αρνητική απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πλήττεται η εμπιστοσύνη που έχουν στην Ένωση. Ας μην ξεχνάμε ότι υφίστανται κυρώσεις, υφίστανται κανόνες που παρεμποδίζουν το να καταψηφιστούν κάποιες προτάσεις στο Συμβούλιο. Θεωρώ ότι υπάρχει τώρα μια καλή ευκαιρία με αυτή τη νέα ιδέα για να ενισχύσουμε την οικονομική διακυβέρνηση. Αλλά θα πρέπει να ευθυγραμμίσουν τη δράση του και τα κράτη-μέλη, όπω ακούσαμε από του προλαλήσαντε. Να μην εφαρμόζονται, ε, εμφανίζονται συγγνώμη, μόνο στο δεύτερο εξάμεινο και τελικά να καλούνται να υλοποιήσουν τα μέτρα που θα έχουν αποφασιστεί στο ευρωπαϊκό εξάμεινο, το πρώτο εξάμεινο. Δεύτερον, η, η, η ενότητα τη νομοθετική διαδικασία Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να το συνεχίσουμε υπό συνθήκε δημοκρατία και διαφάνεια, να μπορούμε να προβλέψουμε τα αποτελέσματα του όπως είπε, υπόθηκε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μην ξεχνάμε ότι προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας. Τι σημαίνει αυτό. Με τις προτάσεις που έκανε τώρα η Task Force δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δημιουργείται προηγούμενο γιατί πρέπει να επαναλαμβάνεται αυτό στις νομοθετικές διαδικασίες που σχετίζονται με τις μεγάλες οικονομικές ε, μεταρρυθμίσεις ε, που οφείλουμε να κάνουμε. Τώρα, αναθεώρηση της συνθήκης της Λισαβόνας. Ε, τόσο λίγο χρόνο μετά από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης. Περ πρόκειται. Ή θέλουμε να δώσουμε ένα καλό νέο, αν θέλετε, σε όλου τους Ευρωπαίους. Αν δεν μπορούμε να το κατοχυρώσουμε αυτό, δεν αξίζει ο κόπο στόχους. Τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να ε, συμβάλλουν ενεργά στην προετοιμασία τη νέα συνθήκη. Ε, Ιδάλω, μην νομίζετε ότι θα ε, παρακάμψουμε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε εν ώψη της έγκριση συνθήκη τη Λισαβόνα και τη συνταγματική συνθήκη. Θα πρέπει να περιοριστούμε στην οικονομική πολιτική. Ναι, μεν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητα πρέπει να γίνει απλουστευμένη αναθεώρηση, με την απλουστευμένη μάλλον διαδικασία αναθεώρηση συνθήκη Λισαβόνα. Δεν προβλέπει προβλέπεται αυτό στη συνθήκη. Ο κύριος ε, Μίλαν Σβέρ τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να μιλήσω ενώπιόν σας στη σημερινή μας συνάντηση. Λυπούμε που δεν παρίστανται πολλοί βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζω στο μέλλον όλες οι πολιτικές ομάδες ε, να αποφασίσουν τι θα γίνει με τις ε, αντιπροσωπείες τους, ε, γιατί είναι ένα γεγονός που μας γεμίζει χαρά αυτή η συνάντηση με τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. όλοι οι φορείς της αγοράς, ξέρετε, δεν πρόκειται να μας μας βοηθήσουν να βγούμε από την κρίση. Θα δώσουν κάποιες προσωρινές ε, απαντήσεις. Ε, στην έκθεση Μόντιδη ε, αναφέρεται ότι υπάρχει σοβαρό χάσμα ανάμεσα σε αυτά που παρέχονται μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ευρώπη και των αναγκών που διαπιστώνονται στην αγορά εργασίας υπάρχει κάτι πλημελές στο εκπαιδευτικό σύστημα, εάν το αποτέλεσμα δηλαδή των προσπαθειών του εκπαιδευτικού συστήματος δεν συνάδει με τις ανάγκες της αγοράς. Ε, μέσα στην έκθεση Μόντι αναφέρεται επίσης ε, ότι ακόμη και αρνητική οικονομική ανάπτυξη Υπάρχουν κάποια στοιχεία που χρειάζονται οι ευρωπαϊκές οικονομίες, αλλά δεν προσφέρονται από κανέναν. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα απ' όλα να φέρουμε σε πέρα σε μία ε, εις βάθος ε, αναθεώρηση των εκπαιδευτικών συστημάτων, μιλάμε για την ε, δευτεροβάθμια εκπαίδευση γενικά, είτε για την επαγγελματική κατάσταση, ή για τη διαδικασία της Μπολόνια, την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα πρέπει να έχουμε μια πιο κρατεή βάση αν ε, θέλουμε η Ευρώπη να έχει τα μέσα που χρειάζεται. Ευχαριστούμε. Ζητώ συγγνώμη ε, και λυπάμαι, αλλά έχει κλείσει ο κατάλογος των ομιλητών. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, γιατί αλλιώς δεν θα ακούσουμε ε, τα μέλη του πάνελ και δεν νομίζω να θέλετε κάτι τέτοιο. Μη μου στέλνετε άλλα ονόματα. Έχει κλείσει ο κατάλογος των ομιλητών. Τελευταίος ομιλητής είναι ο κύριος Κράινερ. Ο κύριος Σέπτσικ από την ε, Τσεχική Γερουσία. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που διοργανώσετε αυτή την εξαιρετικά σημαντική συνεδρίαση. Ούτε κανένα φορέας, ούτε η Κόζακ δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια τέτοια συνεδρίαση. Οι μικτές κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις είναι το η πιο κατάλληλη σκηνή, η το πιο κατάλληλο φόρουμ για να συζητηθούν αυτά τα καυτά ερωτήματα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κρίση αυτή η οποία ξέσπασε μετά την επικύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας και δεδομένου τώρα έχουμε την συνθήκη της Λισαβόνας τα ζητήματα έχουν γίνει πιο καυτά και πιο επίγοντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύω ότι συμπεριφέρθηκε πάρα πολύ καλά στην κρίση αυτή όπως ανέφερε και ο κύριος Ζουαγέ απέφυγε ένα πάρα πολύ σημαντικό κίνδυνο δηλαδή να καταφύγει στον ε, προστατευτισμό. Αυτό το καταφέραμε. Ο κύριος Ζωγέ ήταν ε, ε, ε, τότε, στην, αρμόδιος υπουργό τότε και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη γραμμή που ακολούθησε ως Γάλλος υπουργός. Όσον αφορά την εσωτερική αγορά, ορισμένοι είναι υπέρ μεγαλύτερων ρυθμίσεων, αλλά ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κατεύθυνση των συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι προτιμάτε, περισσότερο ρύθμιση προστατευτισμό ή λιγότερο και απελευθέρωση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Γκέρες Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να πω κάποια πράγματα πρόεδρο. Τώρα αν έχουμε ξεπεράσει ήδη την κρίση αυτό δεν το ξέρουμε αλλά γνωρίζουμε κάτι ξεκάθαρα ότι πρέπει να κάνουμε το παν για να μην επανελειφθεί μια παρόμοια κρίση. Διότι αν επαναληφθεί δεν θα έχουμε πια καμία δυνατότητα να, να ανταπεξέλθουμε επιτυχώς. Άμα δείτε ποια είναι τα συμπεράσματα από την κρίση μέχρι τώρα και τι έχει συμβεί, τότε πιστεύω ότι θα πρέπει να συγχαρούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι ασχολήθηκε αμέσως και με πολύ μεγάλη σοβαρότητα με τα θέματα της αντιμετώπισης της κρίσης και τα θέματα του απαραίτητου ελέγχου και εποπτείας των ε, οικονομικών πτυχών. Πρέπει λοιπόν να το συγχαρούμε. Είναι κρίμα, είναι αλήθεια, που τόσο λίγοι ευρωβουλευτέ είναι παρόντες. Θα μπορούσαμε να είχαμε εμβαθύνει στη συζήτηση, αν ήταν περισσότεροι παρόντες, ίσως την άλλη φορά θα έρθουν περισσότεροι. Τώρα τα συμπεράσματα τα οποία θα πρέπει να συνάγουμε από την κρίση. Πριν από τα συμπεράσματα πρέπει εγώ να ξέρω την απάντηση στο εξή ερώτημα. ποιο πληρώνει τα σπασμένα, τα σπασμένα τα πληρώνουν οι πολίτες οι πολίτες μας. Θα πρέπει λοιπόν να συμμετάσχουν στις ε, λύσεις, ε, στην εξέβρεση λύσεων για τις κρίσεις αυτές, αυτής οι φορείς που τη δημιούργησαν, οι πέτη δηλαδή, δηλαδή αυτοί οι οποίοι έκαναν όλες αυτές τις καταχρηστικές οικονομικές συναλλαγές που χρησιμοποίησαν, προώθησαν και πούλησαν όλα αυτά τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία δημιούργησαν, έδωσαν το έναυσμα για αυτή τη σοβαρή κρίση. Άρα λοιπόν οι υπεύθυνοι, οι υπέτοι πρέπει να βοηθήσουν και να χρηματοδοτήσουν τις απαραίτητες λύσεις. Διαφορετικά ε, δεν θα μπορέσουμε να περιορίσουμε και να κάμψουμε αυτή την τρελή και παράλογη πορεία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Η, η μεγάλη λοιπόν ε, ε, κερδοσκόποι πρέπει να μοιραστούν την ευθύνη των λύσεων και στην Γερμανία εν ώψη της ε, νέας νομοθεσίας ε, για την φορολόγηση των ε, οικονομικών συναλλαγών θα πρέπει να μελετήσουμε όλες τις δυνατότητες συνετής διαχείρισης της Ευρωζώνης και του Ευρώ. Ευχαριστώ. σε πολλές μικτές διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις στις οποίες έχω ήδη συμμετάσχει. Ε, η συμμετοχή ευρωβουλευτών στις προηγούμενες παρόμοιες συνεδριάσεις δεν ήταν ούτε καλύτερη ούτε χειρότερη και η παρουσία ευρωβουλευτών είναι άσχετη με το αν συνεδριάζουν άλλες επιτροπές τις οποίες είναι μέλη. Αυτό το οποίο πρέπει να επιδιώξουμε είναι να έρχονται περισσότεροι. Ίσως ε, θα πρέπει να αλλάξουμε την αντιστοιχεία ομιλητών, να μην είναι δύο από τα Εθνικά Κοινοβούλια και ένας Ευρωβουλευτής, να, αλλάξουμε αυτή την ισορροπία, μπας και τους παρακινήσουμε να έρθουν. Στο θέμα της εναρμόνισης ε, των, της φορολογίας, των φόρων, ε, Βεβαίως, ε, σε μια χώρα όπου η φορολογία είναι χαμηλή, μπορεί μακροπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα να δημιουργήσει μια μεγάλη έλξη κεφαλαίων εν συνεχεία παρακινδυνευμένες καταστάσεις και στο τέλος αυτή η χαμηλή προκλητική φορολόγηση να ζημιώσει όλη την Ευρωζώνη. Εδώ και χρόνια υπάρχει, γίνονται έντονες προσπάθειες εναρμόνισης του, της φορολόγησης των εταιριών πιστεύω ότι προς αυτή την πορεία πρέπει να, αυτή την πορεία πρέπει να ακολουθήσουμε και όχι εν θερμό να αποφασίσουμε απότομες αυξήσεις του φορολογικού συντελεστή, αλλά να επιδιώξουμε την εναρμόνιση της φορολόγησης τουλάχιστον εκεί που μπορούμε στην, ε, στον επιχειρηματικό τομέα, στις εταιρείες, στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία. Δεν είναι εύκολο να ε, ε, εναρμονίσουμε την φορολογία και γι' αυτό δημιουργούνται και πάρα πολλές ε, καταχρήσεις. Εάν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημειωθούν μεγάλες αντι, αντιδράσεις, τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να εναρμονίσουμε ε, και να σταθεροποιήσουμε ε, τα στοιχεία της Ευρωζώνης. Τώρα ποιος πρέπει να πληρώσει τα σπασμένα, αυτοί οι οποίοι εποφελήθηκαν από τις κερδοσκοπικές ενέργειες πρέπει οπωσδήποτε να συμμετάσχουν και να αναλάβουν ισομερώς τις ευθύνες. Ε, φορολογούμε ένα λίτρο γάλα με 5-10% ε, φορολογούμε ένα παλτό που φοράμε με 10% φόρο κατανάλωσης αλλά φορολογούμε ορισμένες μετοχές ή ε, ορισμένες ε, οικονομικές συναλλαγές με συντελεστή μηδέν. Δηλαδή δεν πληρώνεται καθόλου φόρος. Εγώ θα έλεγα ότι τα πράγματα θα έπρεπε να είναι ανάποδα. Ευχαριστώ. Για να ολοκληρώσουμε τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Ντανιέλ Πασκέλ από το Εθνικό Κοινοβούλιο της Γαλλίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Συγγνώμη, έχουμε μία μπλε κάρτα. Σας διακόπτω γι' αυτό το λόγο. Μπορείτε να συστηθείτε κιόλας και να υποβάλλετε το ερώτημά σας προς τον κύριο Κράινερ. Είμαι ο Γιάν Πέτρεσον από τη Σουηδία. Ε, δέχεστε κύριε Κράινερ να απαντήσετε στο ερώτημα του κύριου Πέτρεσον. Βεβαίως, όταν την ακούσω θα απαντήσω. 30 δευτερόλεπτα. Κοιτάξτε, για το φόρο των συναλλαγών των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Έχετε κάποια εμπειρία από χώρα που να έχει εφαρμόσει αυτό το φόρο. Εάν όχι, θα μπορούσα εγώ να σας μιλήσω για τη δική μας εμπειρία. Ε, τη δεκαετία του 80 στη Σουηδία είχαμε ένα τέτοιο φόρο. Για ένα χρόνο κράτησε ε, και μετά εγκατελείφθη το, το πρόγραμμα, το φόρος αυτός. Ναι. Το ξέρω ότι η Σουηδία είχε ένα φόρο επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών και ότι εν συνεχεία καταργήθηκε. Αυτό είχε, είχε σχέση με την αναλογικότητα. Δηλαδή, αν μια χώρα το επέβαλε αυτό, θα έπρεπε και οι άλλες να το επιβάλλουν διαφορετικά. Δεν μπορούσε να το επιβάλλει μόνο αυτό το φόρο μία χώρα και αυτό το κατάλαβε και η Σουηδία πολύ γρήγορα και είπε ότι μόνη μου δεν μπορώ να προχωρήσω, ε, μονομερός δηλαδή. Δηλαδή, ε, γι' αυτό ε, πιστεύω ότι τώρα έχει γίνει ε, κατανοητό ότι χρειάζεται ένα τέτοιος φόρος πια παγκοσμίω και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την έστω σύντομη σουηδική εμπειρία. Ευχαριστώ κύριε Κράιναρ. Για τρία λεπτά ο κύριος Πασκουέλε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, τον Πρόεδρο Λιέ, τον Πρόεδρο των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων της, ε, του Κοινοβουλίου μας εκπροσωπώ εδώ. Χαίρομαι που παρίσταται ο Ζαν Ζουγιέ. Ήταν πολύ ένας διακεκριμένος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και είχα τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του. Νομίζω ότι υπάρχει συνένεση περί των προκλήσεων. Ε, δεν θέλουμε λιγότερη Ευρώπη, περισσότερη Ευρώπη χρειαζόμαστε και έχουμε και, οικονομικά και, πολ... και οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις εσωτερικό επίπεδο οικονομικέ προκλήσεις. Η εσωτερική αγορά δεν έχει ολοκληρωθεί ε, σήμερα. Υφίστανται οξύε ανισότητες ω προς το περιβάλλον, τη φορολογία και την κοινωνική πολιτική και θα πρέπει να τίνουμε προς αυξημένη εναρμόνιση των νομοθετημάτων, των εθνικών νομοθετημάτων ε, ούτως ώστε να έχουμε την ανταγωνιστική θέση που μα αξίζει και να επικρατούν ε, ε, συνθήκες θεμητού ανταγωνισμού. Επίσης, έχουμε σε διεθνές επίπεδο οικονομικές προκλήσεις. Η Ευρώπη δεν έχει επαρκώς κρατεά θέση για να επιβληθεί στην παγκόσμια σκηνή, στον ΚΑΤ, στον ΠΟΕ. Ε, μελλοντικά στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, κατά τη γνώμη μου, η Ευρώπη πρέπει να μιλάει με μία φωνή μόνο ενώπιον των εταίρων της ε, για να μην χρησιμοποιούν αυτές τις ε, διχογνωμίες οι εταίροι της Ένωσης. Βλέπετε τι έγινε με τις διαπραγματεύσεις με την Κίνα. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ενωμένοι, να υπερασπιζόμαστε καλύτερα τα συμφέροντά μας στην παγκόσμια σκηνή εν ώψη της αδύρυτης ανάγκης αμοιβαιότητα στα πλαίσια των εμπορικών διαπραγματεύσεων ω προ όλε τι υπόλοιπε χώρε του κόσμου. Ε, Επίση, έχουμε ένα θεσμικό πλαίσιο που βελτιώθηκε με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, λοιπόν, θα πρέπει να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται η συνθήκη τη Λισαβόνα, αλλά δεν επαρκεί. Ε, η παρά είναι περίπλοκο, εξακολουθεί να είναι υπερβολικά περίπλοκο το σύστημα και ε, βλέπουν πόσα δύναμη η θέση της Ευρώπης στην παγκόσμια σκηνή και ε, μπορούμε να αναρωτηθούμε πόσο μπορεί να δίνει εύκολα απαντήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχύσει την παρουσία της ε, στην παγκόσμια σκηνή θα πρέπει επίσης ε, στο ιστορικό της, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει σαφής καθοδήγηση ε, της εσωτερικής αγοράς. Η Γαλλία και η Γερμανία ζήτησαν οικονομική διακυβέρνηση για την Ευρώπη και προσυπογράφω ε, αυτό το στόχο. Χρειάζεται, είτε μιλάμε για τα οικονομικά είτε για τα πολιτικά ζητήματα, εξάλλου αλληλένδετα είναι και ο κύριος Σούμαν ε, το 1950 στη δήλωσή του το διευκρίνησε αυτό επαρκώς. Χρειαζόμαστε περισσότερο Ευρώπη σε πολιτικό και σε οικονομικό επίπεδο και θα κλείσω έτσι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ολοκληρώθηκε τώρα ο κατάλογος των ομιλητών. Ε, υπερβήκαμε κατά τι το χρόνο, αλλά δεν πειράζει. Θα ακούσουμε τώρα τις απαντήσεις ε, από τον συνάδελφό μας, τον κύριο Ζουγέ. Ακούσα τις παρεμβάσεις ε, των ε, βουλευτών ε, και θα ήθελα να αδράξω την ευκαιρία για να σας ευχαριστήσω για τη δουλειά που έχετε κάνει κατά το εξάμεινο της Γαλλικής Προεδρίας. Καθημερινά συνεργαζόμασταν σχεδόν. Καταβάλλατε υπεράνθρωπη προσπάθεια και σας ευχαριστώ και για τη σημερινή σας παρουσία εδώ. Ο κύριος Ζουγέ, ευχαριστώ Πρόεδρε Ισπανιστή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τα καλά σας λόγια για τη ε, αυροφροσύνη σας. Ε, δεν ξέρω αν τα αξίζω, περνάει στα γαλλικά ο μιλητής. Ε, δεν ξέρω αν αξίζω τα καλά σας λόγια, πάντως σας ευχαριστώ ολόφερμα, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ομαδοποιήσω τις απαντήσεις μου. Υπάρχουν κάποιες που θα αφήσω στον κύριο Μαρτίνες και λιγότερο στην κύριο Ντεχό, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω για την εσωτερική λειτουργία του Κοινοβουλίου. Εδώ είναι θέμα κατευθυντηρίων γραμμών του Κοινοβουλίου. Προφανώς ε, θα αποφύγω το να ε, παρέμβω εγώ και να ε, προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα. Θα ήθελα να κάνω τρεις βασικές παρατηρήσεις σε σχέση με τις παρεμβάσεις σας. Πολλοί και από εσά και χαίρομαι που όλα αυτά διαμείβονται στα πλαίσια της Μικτής ε, κοινοβουλευτική Επιτροπής ε, με σε συνεργασία των Εθνικών Βουλευτών και των Ευρωπαίων Βουλευτών. Ε, το θέμα, αναφέρομαι στο θέμα των δημοσιονομικών μέσων. Ε, δεν έχω ψευδεστήσεις, αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται διάλογος ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια για αυτό το θέμα, διότι ε, ζούμε μία κρίση εμπιστοσύνης ε, και ορισμένες φορές μπορεί να ε, τρέχουμε ψευδεστήσεις, να πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς όμως να έχουμε τα πετούμενα μέσα στη διάθεσή μας. Εάν όμως δεν επαρκούν τα μέσα ή αν δεν κρίνουμε ότι πρέπει να γίνουν έλεγχοι, πρέπει να διορθωθούν κάποιες οικονομίες, πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να το πούμε, πρέπει να επικρατήσει διαφάνεια στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών για αυτά τα ζητήματα. Ε, και μπορούμε να συνδέσουμε αυτά που γίνονται σε επίπεδο προϋπολογισμού της Ένωσης και Οικονομικής Πολιτικής Ένωσης ε, και να τα συνδυάσουμε ε, με την αλληλέγγυα χρήση κάποιων μέσων στα πλαίσια κάποιων πολιτικών, όπως είπε ένα συνάδελφος. Έχουμε τους εταίρους, έχουμε τις αγορές και πρέπει να συνεργαστούμε με όλους αυτούς τους συνομιλητές για να δούμε ποια οικονομική πολιτική θα ακολουθήσουμε. Ο κύριο Καρέ, επίσης είπε κάτι σωστό. Είπε τίποτα ότι θα ήταν χειρότερο από το να έχουμε στρατηγικέ χωρίς χρηματοδότηση. Κοιτάξτε, οι αγορές είναι περίπλοκα μέσα. Ε, ορισμένες φορές το υπερβολικά περίπλοκα, αλλά μην μπερδεύεστε, τα πράγματα είναι απλά. Ε, κάθε στρατηγική θέλει και τη χρηματοδότησή της. ε, όπως λειτουργούν τα πράγματα κανονικά δεν υπάρχει καμία διαφορά ως προς τον τρόπο λειτουργία των θεσμικών οργάνων. Ε, κάθε στρατηγική χρειάζεται χρηματοδότηση. Και σε διαβούλευση και με όλους τους εταίρους μπορεί να βρεθεί αυτή η χρηματοδότηση. Δεύτερη παρατήρηση, και ζητώ συγγνώμη που θα εκφραστώ έτσι, ε, πρέπει να ακούσουμε τις αγορές να αφουγκραστούμε τις ε, αγορές. Είναι εύστοχα τα ερωτήματα που θέτουν οι αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο είδη ερωτημάτων που θέσατε και εσείς εξάλλου προέρχονται από τις αγορές. Πρώτον, η σύνδεση ανάμεσα στα βραχυπρόθεσμα και τα μεσοπρόθεσμα μέτρα. Κάποιοι επέμειναν για τη σημασία τη βιώσιμη ανάπτυξη, για τη χρηματοδότηση έρευνα και τη ανάπτυξη. Ναι, ναι. Ε, αυτό πρέπει να γίνει στα πλαίσια τη πολιτική 2020. Ναι, ναι, όλα αυτά ναι. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να απαντήσουμε και στι βράχυπρόθεσμε προκλήσει. Να δώσουμε μια απάντηση στα προβλήματα των προσαρμογών. Ε, νομισματικών και άλλων στα προβλήματα της ε, οικονομικής διακυβέρνησης της ζώνης ευρώ για να διαπιστώσουμε αν αυτά τα προβλήματα, μάλλον σε τι έγκυται αυτά τα προβλήματα. Θα πρέπει να δοθούν εθνικές απαντήσεις με μέτρα ε, προσαρμογής, δημοσιονομικής προσαρμογής, με μέτρα που προβλέπονται ήδη στο νομισματικό πεδίο και πώς να κατεχειρώσουμε τη συνοχή ανάμεσα στα επιμέρους μέτρα και επίσης το ζήτημα της διαφάνειας και τις σχέσεις ε, που υπά... το σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στα διάφορα κρατικά δάνεια. Όλα αυτά τα αρετήματα θα πρέπει να τα απαντήσουμε ε, Επίση, οι βραχυπρόθεσμε απαντήσεις που θα δώσουμε στις αγορές θα πρέπει να συνδυαστούν με τη μέσοπρόθεσμη στρατηγική μας. Αυτό αναφέρθηκε και οφείλουμε να γνωρίζουμε αν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να αναλάβει δέσμευση προς μια σαφέστερη πολιτική ε, είτε για το δανεισμό σε επίπεδο ένωση είτε για τη διαχείριση των χρεών πάλι σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή αν δεν το επιθυμούμε αυτό, τέλο να πούμε προς τα πού θα οδεύσουμε για τον φορολογικό ανταγωνισμό, ε, για τον ε, νομισματικό ανταγωνισμό. Το αναφέρατε εσείς, ε, αναρωτιούνται οι αγορές, αναρωτιούνται και οι εταίροι μας. υπάρχει αυτή η σχέση ανάμεσα στις επιτακτικές ανάγκες ε, ε, της βραχυπρόθεσμης και της ε, μέσοπρόθεσμης. επίσης για την οικονομική πολιτική, και αυτό το ανέφεραν πολλοί συνάδελφοι, ο κ. Βαμπεμέλ, παραδείγματος χάρη, επανήλθε σε αυτό το θέμα και άλλοι βέβαια για τον συνδυασμό των, ε, των πολιτικών ε, προσαρμογής και λιτότητας σε ορισμένες περιπτώσεις και ε, το συνδυασμό τους λοιπόν με τις αναπτυξιακές πολιτικές. Ε, ζητούμε περισσότερη λιτότητα πάντα. Όχι, αναρωτιόμαστε ποια είναι η ακολουθητέα στρατηγική. Πώ θα επιτύχουμε την καλή ισορροπία ανάμεσα στην υποστήριξη τη οικονομική δραστηριότητα και των προσπαθειών που πρέπει να γίνουν για το χρηματοπιστωτικό ε, και ε, για τη χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική προσαρμογή. Και πρέπει να είναι σαφέστατε οι απαντήσει μα σε σχέση με τι προσδοκίε των επενδυτών. Δεν είναι από τι ίσονε δυσκολίε αυτή που, στην οποία αναφέρομαι. Ο κύριο Ζολιμέρ το τόνισε εξάλλου και άλλοι. Ε, πέρα από την υπέρβαση της κρίσης ε, που επιτύχαμε εν μέρη, μην ξεχνάμε ότι ε, ακόμη την βιώνουμε και κυρίως την υποτροπή πρέπει να αποφύγουμε. Οι στρατηγικές μας θα πρέπει να συντονιστούν και να οριοθετηθούν επακριβώς για τις ε, διάφορες δόσεις όλων των συστατικών, ε, δηλαδή λιτότητα από τη μία και ανάπτυξη από την άλλη. Ε, Γιατί τώρα η τρίτη μου παρατήρηση για τι αγορέ. Είπαμε πρέπει να ακούμε τι αγορέ. Ναι, ταυτόχρονα όμω να εποπτεύουμε, να επιβάλλουμε κυρώσει ε, και να καταπολεμούμε τι τρέλε των αγορών. Ε, να, όταν υπερθερμαίνονται να τι επαναφέρουμε στη σωστή θερμοκρασία, όπω είπαν πολλοί συνάδελφοι. Και από αυτού πρέπει να είμαστε σαφεί. Όπως ο κύριος Δεμέλ, θα νομίζω πρέπει να κάνουμε και εμείς μια αξιολόγηση των ε, φιλελευθέρων πολιτικών που ακολουθήθηκαν σε διάφορες αγορές. Ε, δεν πρέπει να φοβόμαστε. Πρέπει να καταπολεμήσουμε την υπερβολική νευρικότητα των αγορών, ε, την υπερβολική αδιαφάνεια κάποιων άλλων. Πρέπει να είμαστε σαφέστατοι. Η Ευρώπη πρέπει να λειτουργήσει με στένος και πυγμή. Για να καταπολεμήσουμε την υπερθέρμανση των αγορών, τι πρέπει να κάνουμε. Ναι, να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά το θέμα της, ε, του φόρου των ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ε, και είναι ευκταίο σε ορισμένες περιπτώσεις να επιβληθεί ένας τέτοιος φόρος τώρα αν προκύψει ότι μπορώ, πρέπει και πρέπει, μπορούμε να το κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα το κάνουμε. Πρέπει να είμαστε υποδειγματικοί. Φυσικά προφαν... είναι προφανέ ότι είναι καλύτερο να συμβεί αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά δεν θα πρέπει να καταλήψουμε την ιδέα γι' αυτό το λόγο, να το συζητήσουμε με άλλου εταίρου και να δούμε αν ενδείκνυται να εφαρμοστεί ένα τέτοιο φόρο και τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπω και σε άλλου τομεί. Γιατί νομοθετήσαμε σε τόσου διαφορετικού τομεί. Ε, δεν καταλαβαίνω γιατί ε, στον τομέα των αγορών, των χρηματοπιστωτικών αγορών, αγορών να αποφεύγουμε μια τέτοιου είδου ρύθμιση, θα, να αποφύγουμε την υπερθέρμανση των αγορών, να καταπολεμήσουμε τι τρέλε των αγορών, τι υπερβολέ των αγορών, να, να επιβληθεί η Ευρώπη. Δεν ναι, αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη ΣΥΠΑ, άρα είναι λογικό να δίνει και διαφορετικέ απαντήσει ε, ε, σε σχέση ε, και με αυτά που πρέπει να κάνει ε, για, στη σχέση της με τους εταίρους, άλλους εταίρους, πέρα από ό,τι είπα. Ε, τώρα, συνεχίζοντας να απαντώ στις ερωτήσεις, θα περάσω ειδικότερε παρατηρήσεις. Χρειάζεται καλύτερος οικονομικός συντονισμός και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα, ε, βρίσκουμε βραχυπρόθεσμες απαντήσεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Είδατε όμως τα δύο τελευταία χρόνια, βρήκαμε απαντήσεις στο ιστορικό της Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν έχουμε τόσο διαφορετικές απόψεις από αυτές που προβάλλουμε στη σχέση μας με τον υπόλοιπο κόσμο. Βέβαια, ακόμη θα πρέπει να σημειωθεί πρόοδος για να συντονίσουμε τις θέσεις μας. Και κλείνοντας, ε, θα ήθελα να κάνω την εξή παρατήρηση. Ξέρουμε πως ε, δεν μπορούμε να υπερβούμε τον ορίζοντα Ευρώπη. Ε, δηλαδή τι εννοώ, είναι αναπόφευκτο να έχουμε περισσο... όλα και περισσότερη Ευρώπη. Το είπατε και εσείς, χρειαζόμαστε περισσότερη αλληλεγγύη στο εσωτερικό της Ένωσης και ε, κυρίως σε σχέση με τα βασικότερα θύματα σε εισαγωγικά της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Όμως δεν πρέπει να τρέφουμε και ψευδεστήσεις. Χρειαζόμαστε την αλληλεγγύη, αλλά ταυτόχρονα ε, και την ορατότητα. Την, ε, πρέπει δηλαδή να γίνονται όλα κατανόητα, αντιληπτά από την κοινή γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τελευταία δύο χρόνια. Ε, τι βλέπουμε, ότι ενισχύεται η αλληλεγγύη, όμω δεν ενισχύεται αντίστοιχα και η εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτε στα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι μια πρόκληση ε, που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε αυτή την τόσο δυσχερή περίοδο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ζουγέ για το όσα μας είπατε. Τώρα θα έχουμε τις συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας που σίγουρα θα εμπνευστούν και από τη δικιά σας παρουσίαση. Τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα θα χωριστούμε σε τρεις ομάδες. Τρεις ομάδες εργασίας. Η πρώτη ομάδα εργασίας που έχει ως τίτλο τι είδους ανάπτυξη και τι είδους απασχόληση θέλουμε για την αυριανή Ευρώπη θα λάβει χώρα εδώ. Είναι ο φίλος και συνάδελφος Μιγγέλ Πόρτας Ευρωβουλευτής που θα προεδρεύσει μαζί με την κυρία Μαρία Ρένα που είναι από τη Βελγική Γερουσία. Ο εισηγητής της ομάδας αυτής της εργασίας θα είναι ο κύριος Μπρούνο Τάιμπενς που είναι Βέλγος βουλευτής από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ενώ η κυρία Ρένα είναι από τη Γερουσία. Η ομάδα αυτή θα εργαστεί εδώ. Ενώ οι υπόλοιποι πρέπει να μετακινηθούμε. Η ομάδα εργασίας 2 που λέει τι είδους ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση θέλουμε θα συνεδριάσει στην αίθουσα 3C050 στον τρίτο όροφο του ίδιου κτίριου. Δηλαδή στον ίδιο όροφο θα βγείτε έξω και είναι απέναντι θα συνεδριάσει ο γνώσιν συμπρόεδρο εδώ, ο συνάδελφος Χέρμαν Τεκρό. Που είναι από το Βελικό Κοινοβούλιο, την Βουλή των Αντιπροσώπων, το Άγιο Πνεύμα κλπ. κλπ λέει ο Πρόεδρος. Θα συμπροεδρεύσει ο συνάδελφός μας Χωσέ Μανουέλ Γκαρθία Μαργάγιο Μαρφίλ. Η τρίτη ομάδα θα ασχοληθεί με το πώς να ολοκληρωθεί, πώς να τελειώσει η ενιαία αγορά. Θα συνεδριάσει στην αίθουσα 1α002. Α, συγγνώμη. Όχι. Μαζί με τον κύριο Ντεκρό θα είναι ο κύριος Γκοζές, λέει ο πρόεδρος. Και η τρίτη ομάδα, στον πρώτο όροφο αυτού του κτηρίου, στην αίθουσα 1α002, θα προεδρεύσουν ο κύριος Μάλκομ Χάρμπορ, ο Ευρωβουλευτής, και ο κύριος Λάγιος Μίλε από την Ουγγρική Βουλή. Και η συγκητής εκεί θα είναι ο κύριος Γιώργη Βιλαγιωάννα, που είναι μέλος της Ισπανικής Γερουσίας. Τι άλλα σχόλια έχω να σας πω. Σας είπα πώς θα πάτε στις διάφορες αίθουσες δεν νομίζω ότι θα χαθείτε. Αν και πάντα είναι εύκολο να χαθεί κανείς σε αυτό το λαβύρινθο που βρισκόμαστε. Πάντως θέλω να σας υπενθυμίσω ότι οι ομάδες εργασίας πρέπει να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους στις 7. Οι εισηγητές από τις τρεις ομάδες εργασίας θα παρουσιάσουν καλύτερα γραπτά και στα αγγλικά ή στα γαλλικά τα συμπεράσματά τους αύριο το πρωί. Έτσι ώστε εφόσον τα έχουμε και γραπτά μπορούμε να τα μοιράσουμε και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Κατά τα άλλα θα το ξέρετε βέβαια, αλλά σας το λέω και εγώ ότι στις 7 και 4 υπάρχει κοκτέιλ που προβλέπετε και δείπνο στη συνέχεια. Υπό την προεδρία του κυρίου Γέρση Μπούζεκ έχουμε την τιμή δηλαδή να μας καλεί στον χώρο Γεγουντή Μενούχιν που είναι στο κτίριο αυτό αλλά στον πρώτο όροφο. Αυτά. Τα έχετε και στα έγγραφα τα οποία σας έχουν μοιραστεί αναφέρονται πληροφορίες αυτές. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά τον συνάδελφο Ντεκρό που με βοήθησε εδώ στην Προεδρία και με συνόδευσε σε αυτήν. Εύχομαι καρποφόρες εργασίες στις ομάδες εργασιών και θα τα πούμε αργότερα όλοι μαζί. Και εκεί θα μας δοθεί και ευκαιρία να γνωριστούμε και καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ.